Ωραία, ας ξεκινήσουμε λοιπόν ε, σιγά σιγά με κάποιες ανακοινώσεις. Λοιπόν, κοιτώντα την ημερήσια ε, διάταξη υπάρχουν ε, δύο σημεία ένα που αφορά το σχολιασμό του δεύτερου τριμερούς ε, διαλόγου για την πρόταση προσβασιμότητας ε, στις ιστοσελίδες ε, του δημόσιου τομέα και ξέρω ότι πολλοί από εσάς εδώ στην αίθουσα ενδιαφέρεστε για ζητήματα προσβασιμότητας ωστόσο αυτή η συζήτηση θα γίνει μετά τις 4 και επίσης ο σχολιασμός του τριμερούς διαλόγου για τις ε, ιατρικές συσκευές και τις in vitro ιατρικές συσκευές. Ο Ντίσης για την πρώτη και Ρόζενχοφ για τον δεύτερο θα μας μιλήσουν. Αναβάλουμε την εξέταση των τροπολογιών ε, για τους μη δασμολογικούς φραγμούς στην ενιαία αγορά, τη σχετική έκθεση, επειδή υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις ε, στην επίτευξη των συμβιβασμών λόγω καθυστερήσεων συναντήσει την περασμένη εβδομάδα. Δεν είναι τίποτα περίεργο, απλά μια κανονική καθυστέρηση. Λοιπόν, με μεγάλη μας τιμή έχουμε εδώ μαζί μας ε, τον ε, Επίτροπο Γύρκη Κατάινεν, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Αρμόδιο για την απασχόληση, την ανάπτυξη της επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα. Όλα αυτά βρίσκονται στον πυρήνα της ενιαίας αγοράς. Ευχαριστούμε λοιπόν που ήρθατε να μας μιλήσετε στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς ε, και Προστασίας των Καταναλωτών. Υπενθυμίζω πάντα ότι είμαστε και Εσωτερικής Αγοράς Επιτροπή. Να το υπενθυμίσετε και στους συναδέλφους σας ε, στην ε, Επιτροπή. Θα ακούσουμε τον κύριο Επίτροπο και τον κύριο Αντιπρόεδρο και μετά θα ακολουθήσει μια σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Είναι πολύ καλή ευκαιρία σήμερα να δούμε την πρόοδο ε, στα θέματα αυτά Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ε, για τα τεκτενόμενα και το που έχουμε φτάσει για τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την ενιαία αγορά και ειδικότερα την απασχολησιμότητα, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα. Δεν θα μπορέσω να καλύψω όλες τις δράσεις μας, ε, οπότε θα εστιαστώ σε κάποια βασικά σημεία που παίζουν ρόλο κλειδί και που, στο στόχους τους δικούς μας και που είναι σημαντικά για την Επιτροπή σας. Θα σας κάνω πρώτα απ' όλα μια ενημέρωση για το που βρισκόμαστε με το επενδυτικό σχέδιο που όπως γνωρίζετε με έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες. Μετά θα πω δύο λόγια για την τρέξουσα κατάσταση όσον αφορά την υλοποίηση της στρατηγικής της ενιαίας αγοράς που απασχολεί ιδιαίτερα την Επιτροπή αυτή. Τα ζητήματα φυσικά της ενιαίας αγοράς συμβαδίζουν με το θεματολογιό μας για βελτίωση της νομοθεσίας στο οποίο θα αναφερθώ στο τέλος της ομιλίας μου και μετά ευχαριστώ να ακολουθήσει ένας διάλογος να απαντήσω στις ερωτήσεις σας αν να ακούσω και τα σχόλια και τις ιδέες που έχετε για τα διάφορα ζητήματα. Επενδυτικό σχέδιο λοιπόν πρώτα απ' όλα. Μέχρι στιγμή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει εγκρίνει 56 προγράμματα προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΦΣΥ. Αυτό αντιστοιχεί σε ποσό επενδυτικό 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ. 56 λοιπόν προγράμματα ύψους 7,2 δις. Περισσότερα προγράμματα ακόμη ε, συνεχίζουν να επιλέγονται κάθε μήνα βάσει της μέχρι στιγμής προόδρου. Ε, έχουμε έργα που αφορούν την ενεργειακή απόδοση και άλλες επενδύσεις που βοηθούν σε ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές διευθυντήτου του άνθρακα. Άλλα προγράμματα περιλαμβάνουν έρευνα και ανάπτυξη, ε, βιομηχανική καινοτομία, υποδομέ για την κοινωνία, μεταφορέ αλλά και πρόσβαση σε χρηματοδότηση για μικρομεσαίε επιχειρήσει. Το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο, το EIF, ε, έχει συνάψει πάνω από 150 συμφωνίε ε, σύναψη μικρομεσαίων επιχειρήσεων με συνολική χρηματοδότηση 3 1,4 δις και περίπου 120.000 ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις αναμένεται να υποφεληθούν αυτές τις χρηματοδότησες Μαζί όλες αυτές οι δράσεις θα οδηγήσουν πιστεύουμε σε συνολικές επενδύσεις κοντά στα 76 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το αποτέλεσμα λοιπόν του πρώτου μήνου. 76 δισεκατομμύρια ευρώ προς ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τη χρηματοδότησή τους και τη χρηματοδότηση προγραμμάτων. 22 κρατημέλη μέχρι στιγμή έχουν αποφεληθεί από το ΕΦΣΥ συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μικρών οικονομιών όπως η Σλοβενία, η Εστονία, η Βουλγαρία και η Κροατία. Η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία είναι οι ηγέτιδες χώρε του Ηνωμένου Βασίλειου ανάλογα με το αν μετράμε τον αριθμό των προγραμμάτων ή τα χρήματα. Ε, είναι αριθμός ένα ή δύο. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Δεν θυμάμαι με ποιον υπολογισμό το νούμερο Βασίλειο είναι η πρώτη χώρα, αλλά ε, η Γαλλία και η νούμερο Βασίλειο είναι οι πρώτες χώρες. Τώρα, ε, όσοι προωθούν ε, προγράμματα συνεργασίας ιδιωτικού δημόσιου τομέα μπορούν να ζητήσουν αρρωγή από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και αργότερα την Άνοιξη θα ξεκινήσουμε την πύλη των Ευρωπαϊκών Επενδύσεων ε, ώστε να διαφημίζουν εκεί τα προγράμματά τους οι διάφοροι ε, όσοι προωθούν τέτοια προγράμματα ε, για επενδυτές. Στις 22 Φεβρουαρίου οι Κομισιόν και ε, δημοσίευσαν ένα έγγραφο ώστε να βοηθήσουν τις τοπικές αρχές και τους υποστήκτες των έργων να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες αξιοποίηση αυτών των κονδύλιων. Αυτά τα δύο εργαλεία έχουν σχεδιαστεί με διαφορετικό αλλά συμπληρωματικό τρόπο. βάσει λογικού σχεδιασμού και ε, του νομοθετικού πλαισίου ενισχύουν ε, ε, το ένα το άλλο και συμπληρώνονται από διάφορες πολιτικές μας έρευνας και ανάπτυξης. Το Horizon 2020 αποσκοπεί σε δημιουργία μιας γνωσιακής βάσης βασισμένης στην αριστεία και σε ένα περιβάλλον το οποίο θα οδηγήσει σε καινοτομία στην Ευρώπη. Καινοτομία ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική ευμάρεια, η ασφάλεια, η ποιότητα διαβίωσης ε, και ποιότητα του περιβάλλοντος ε, σήμερα και για το μέλλον. Το Horizon 2020 παρέχει ήδη αποτελέσματα. Έχουμε ήδη υπογράψει 7.200 ε, συμφωνίες με συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους 12,6 δισεκατομμύριων ευρώ προς 31.000 συμμετέχοντες. Αυτό συμπεριλαμβάνει πάνω από 1.300 ε, χορηγίες, συμφωνίες χορηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης η Κομισιόν είναι πολύ φιλόδοξη για την άρση των συγκεκριμένων ρυθμιστικών φραγμών προς τις επενδύσεις και να δημιουργήσει ένα καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον. Εξετάζουμε τις επόμενες προκλήσεις ε, για τις επενδύσεις που βιώνουν τα κράτη-μέλη. Στις 26 Νοεμβρίου του 2015 υιοθετήσαμε την ετήσια έρευνα που περιλαμβάνει δελτία χωρών όπου περιγράφονται οι φραγμοί για τις επενδύσεις σε κάθε κράτος μέλος. Ήδη η Κομισιόν έχει ξεκινήσει την ε, κοινή αγορά κεφαλαίων, την ε, Ένωση των Κεφαλαίων και την ε, Ενεργειακή Ένωση και αυτές θα δημιουργήσουν ένα καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον για τους επενδυτές. Αργότερα την Άνοιξη θα υιοθετήσουμε επίσης και το θεματολόγιο για τις δεξιότητες, το Skills Agenda η περαιτέρω ενίσχυση και εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στην πρώτη θέση του θεματολογίου μας και πρέπει να άρουμε τους περιορισμούς και τα εμπόδια για επαγγελματίες και για επιχειρήσεις. Η ενιαία αγορά πρέπει να ακολουθεί το πνεύμα των καιρών, ενθαρρύνοντας τις επενδύσεις και τους νέους επιχειρηματίες, καλωσόζοντάς τους στην ενιαία αγορά. Θέλουμε να αναπτύξουμε ένα ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη συνεργατική οικονομία, ώστε να ενθαρρύνουμε την αναπτύξη νέων καινοτόμων υπηρεσιών, χωρίς να ευνοούμε κάποιες επιχειρήσεις περισσότερο από άλλες. Θέλουμε επίσης να εισάγουμε ε, τα μέτρα για τις υπηρεσίες ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών να μπορούν εύκολα να συμμορφώνονται με τις ε, διάφορες απαιτήσεις σε περίπτωση συναλλαγών με άλλα κράτη-μέλη. Θέλουμε να, επίσης να εναρμονίσουμε ορισμένες απαιτήσει σε τομείς προτεραιότητας που, όπου παρατηρούνται χαμηλές επιδόσεις όσων, δηλαδή μιλάμε τώρα για συγκεκριμένες επιχειρήσεις και συγκεκριμένες ε, υπηρεσίες. Θέλουμε να βελτιώσουμε το ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης με προενεργό ε, συμμετοχή και τη συμμετοχή των, ε, της κοινωνίας των πολιτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όλες ε, αυτές οι προτάσεις θα βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα συμπληρώσουν και άλλα μέτρα τα οποία εστιάζονται στη μείωση της γραφειοκρατίας και την πρόσβαση σε επενδύσεις. μέσω ενός επενδυτικού σχεδίου και για τα venture capitals θα βοηθήσουμε την πρόωθηση των οφειών επιχειρήσεων εκ των οποίων μόνο 60% ε, ε, επιβιώνουν σε διάρκεια τριών ετών. Θέλουμε επίσης να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες ΦΠΑ ώστε οι επιχειρηματίες να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία μέσω των νέων κανόνων περιφερειακότητας και θα ξεκινήσουμε και μια πρωτοβουλία για τις νεοφύης επιχειρήσεις ώστε να καταλάβουμε καλύτερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να βοηθήσουμε να μειωθούν οι απαιτήσει συμμόρφωση. Η στρατηγική για την ενιαία αγορά εστιάζεται επίση στην επιβολή του νόμου και στη συμμόρφωση θα δώσουμε συγκεκριμένα εργαλεία για αυτού του σκοπού και θέλουμε να εισάγουμε και ένα εργαλείο πληροφοριών αγορά για την καλύτερη συλλογή πληροφοριών. Επίση, ε, θέλουμε να μεταρρυθμίσουμε ε, τη διαδικασία ειδοποίηση σε περίπτωση υπηρεσιών. Ε, η Κομισιόν παρουσίασε ένα πρώτο σύνολο μέτρων για τα πνευματικά δικαιώματα και τα ψηφιακές συμβάσεις το Δεκέμβριο. Όλο και περισσότερε προτάσεις για τις ψηφιακές τεχνολογίες ε, αναμένονται πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Σε όλου αυτού τους τομείς η προστασία των καταναλωτών ε, έχει προτεραιότητα. και λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις προσπάθειες ε, αξιοποίησης των πλήρων δυνατοτήτων της ενιαία αγορά. Λόγω των μεγάλων προσπαθειών που καταβλήθηκαν για τι συμφωνίε του Παρισιού πρέπει τώρα να δούμε τι θα κάνουμε ω επόμενα βήματα. Προωθούμε το σχέδιο δράση για την κυκλική οικονομία του περασμένου Δεκεμβρίου και καταβάλουμε προσπάθειε για μια αηφόρο ε, ε, ε ανάπτυξη ε, και βάση των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη των ΗΠΑ. Η ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου επίση έχει μεγάλη προτεραιότητα για το 2016 θα μας βοηθήσει να προσαρμόσουμε τις δαπάνες μας ε, ε, βάσει των πολιτικών προτεραιοτήτων. Αυτή την εβδομάδα η Κομισιόν θα εκδώσει μια ανακοίνωση με τα βήματα που θα ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να βελτιστοποιηθούν τα εργαλεία πολιτικής ε, στον τομέα της χαλιβουργίας και για την υποστήριξη της χαλιβουργίας στο μέλλον της. Τώρα, κάποια πράγματα για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Παράλληλα με το θεματολόγιο για βελτίωση της νομοθεσίας, ε, η Κομισιόν προσπαθεί να απλουστεύσει το νομικό πλαίσιο και να μειώσει το διοικητικό άκθος σε ολόκληρη την ενιαία αγορά. Θέλουμε να προωθήσουμε κανονισμούς ε, που να άρουν εμπόδια για την ανάπτυξη, να ελαχιστοποιούν τα κόστη, να δίνουν ευκαιρίες και να διασφαλίζουν ότι η ανάπτυξη θα είναι ε, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη. Γι' αυτό το σκοπό η Κομισιόν θέλει να εστιαστεί σε καλά θεμελιωμένες ε, και ε, πρωτοβουλίες που περιγράφονται σωστά και που θα βασίζονται σε αποτελέσματα και σε παρελθούς εμπειρίες τηρώντας τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Το πακέτο λοιπόν Better Regulation θα επιχειρήσει αυτές τις αλλαγές. Το Better Regulation, η βελτίωση της νομοθεσίας είναι κοινή ευθύνη. Όλα τα θεσμικά όργανα και όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να τηρούν τις αρχές του. Κυρία Πρόεδρε, συνολικά ο διαρθρωμένος μας διάλογος λειτουργεί καλά καθώς προχωράμε προς την εκπλήρωση του προγράμματος Κομισιόν για το 2016 μέσω συντονισμένων συναντήσεων μεταξύ της ε, ε, Επιτροπή Διασκέψη των Προέδρων ε, ε, την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο και τη Κομισιόν. Οι προκλήσεις που έχουμε είναι τεράστιες. Τρομοκρατικές επιθέσεις, η πολύ αργή ανάκαμψη της οικονομίας, οι κλιματικές αλλαγές, η προσφυγική κρίση και οι μεταναστευτικές πιέσεις στα εξωτερικά μας σύνορα και η αίσθηση ανασφάλεια εντό τη γειτονία μα. Όλες αυτές οι προκλήσεις απαιτούν την ανάληψη αποφασιστικής δράσης με αλληλεγγύη και ευθύνη. με διατήρηση του Ηνωμένου Βασιλείου ως σημαντικού παίκτη εδώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ε, συνεργαστούμε όλοι για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να στρώσουμε το δρόμο για να βιώσουμε το πιο ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό μέλλον. Περιμένω με ανυπομονησία το διάλογο μεταξύ μας για να ακούσω τις ιδέες σας, τις απόψεις σας ε, για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχω ανοίξει τον κατάλογο μιλητών, οπότε αν δεν μου έχετε δώσει ακόμα το όνομά σας, μπορείτε να το κάνετε τώρα. Λοιπόν, να καλωσορίσω την κυρία τον κύριο Λότεγκαρτ Μόρτιν. Καλωσορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθιστάτε τον κύριο, την κυρία Τορνές, της οποίας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο της ρόλο στην κυβέρνηση. Καλωσορίσατε λοιπόν στην ε, Επιτροπή ε, Προστασίας των Καταναλωτών και Εσωτερικής Αγοράς. Είναι δύσκολο το έργο μας εδώ. Λοιπόν, να σας πω ποιος έχω στον κατάλογο μιλητών. Στον Κάθριν Νίκολα Ντάνη, Κασιάρη, Άβεν Στέφανιτς, Άντολτ, Φάνος, Τζούλια, Ρέιντα. Take them from in the order of, of groups. So I'm going to... Rosa, did you want to speak first? Θέλετε τον λόγο Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ που βρεθήκατε εδώ και σας ευχαριστώ και για την ε, παρουσίαση. Σας ευχαριστώ λοιπόν που είστε εδώ. Και εγώ πιστεύω, όπως και οι περισσότεροι συνάδελφοι, ότι πρέπει να συνεργαζόμαστε ε, πιο στενά και να ανταλλάσσουμε απόψεις συχνότερα. Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι θα ήθελα να μου πείτε τι έχετε κάνει όσον αφορά την απλούστευση που αναφέρατε. Έχετε λάβει ήδη κάποιες δράσεις, έχετε αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες, κάποια αποτελέσματα. Κάθριν Στάιλερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Πίτροπο που είστε εδώ. Νομίζω ότι η περιγραφή σας για τα 56 προγράμματα και για το EFSI ε, είναι ευπρόσδεκτα. Θα ήθελα να μιλήσω για το θεματολόγιο για τις δεξιότητες. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πάνω από 900.000 ε, θέσεις εργασίας που θα χρειαστούν ε, έως το 2020 συγκεκριμένες δεξιότητες οπότε μπορείτε να μας πείτε εσείς ποιο είναι το όρομά σας γιατί εμείς δεν θέλουμε να διευρυνθεί υπερβολικά αυτή το, το ψηφιακό χάσμα που υπάρχει και ε, μπορούμε δηλαδή υπάρχει ένα τεράστιο, ένα τεράστιο εύρος δεξιοτήτων που χρειάζεται να αποκτήσουν οι άνθρωποι και αν θέλουμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες της ενιαίας αγοράς πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτό το θέμα. Κάτι άλλο για τις θέσεις εργασίας και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, εγώ ε, ε, πρόσφατα ασχολήθηκα με το ζήτημα των ιστοσελίδων και των μικρών επιχειρήσεων ε, και την δυνατότητα της δυνατότητες των μικρών επιχειρήσεων να εμπορεύονται τα ε, προϊόντα τους μέσω ιστοσελίδων. Ήθελα να το τονίσω αυτό και για να πω και κάτι για το τελικό σας σχόλιο για την συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Πιστεύω ότι και εσείς πιστεύετε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να, παραμένει, να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκατό μέρες απομένουν ε, έως το δημοψήφισμα. Από τους μεγαλύτερους ωφελημένους της ενιαίας αγοράς είναι το Ηνωμένο ε, Βασίλειο. Ε, τα πανεπιστήμια μας ωφελούνται από τον ορίζοντα 2020, τι θα συμβεί αν βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, εγώ ανησυχώ γιατί σε κάθε περίπτωση θέλω η χώρα μου να ωφελείται από όλα αυτά που περιγράψατε. Ε, ήθελα να το πω και αυτό μιας και η προηγούμενη ομιλήτρια ήταν πολύ πιο σύντομη. Λοιπόν, να ε, επισπεύσουμε τη συζήτηση γιατί υποσχέθηκα στην προηγούμενη συνάντηση των συντονιστών ότι θα τηρώ το χρόνο με αυστηρότητα. Λοιπόν, έχουμε 10 άτομα, 11 στον κατάλογο ομιλητών και ο καθένας θα έχει ένα-δυο λεπτά. Θα σας διακόπτω όμως αν τα ε, ε, υπερβαίνετε. Dan Dalton. Ευχαριστώ κύριε Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, χάρηκα που σας άκουσα να μιλάτε για την καλύτερη νομοθεσία και συμφωνούμε. Το πρόβλημα είναι ότι η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική, γιατί είναι πολύ απλό να μιλούμε για την απλούστευση και την καλύτερη νομοθεσία, αλλά πολύ συχνά στην πράξη συμβαίνει το αντίθετο. Για παράδειγμα, στα, στην ε, νέα νομοθεσία για τα τελωνία, Έγινε ακριβώς αυτό τελικά. Προκλήθηκαν πολύ μεγαλύτερες ε, επιβαρύνσεις για τις επιχειρήσεις γραφειοκρατικού χαρακτήρα και τελικά χρειαζόμαστε κατεξουδότηση πράξη για να λύσουμε τα προβλήματα. Το ερώτημά μου είναι πώς μπορούμε να επιτύχουμε αυτό το στόχο γιατί ε, συμβαίνει αυτό τελικά όταν προσπαθούμε να ε, επιτύχουμε καλύτερη νομοθεσία. Για τους μη δασμολογικούς ε, φραγμούς πολλές μεσαίες επιχειρήσεις μου λένε ότι είναι πολύ να, κάνουν, να έχουν εμπορικές συναλλαγές με τον Καναδά και τις ΗΠΑ παρά με τη Γερμανία και την ε, Γαλλία. Ε, γιατί υπάρχουν όλοι αυτοί οι μη διασμολογικοί φραγμοί. Εσείς λοιπόν θα υποστηρίζατε να συντάξει η Κομισιόν μια ετήσια έκθεση σε σχέση με την κατάργηση των μη δασμολογικών φραγμών για να εντοπιστούν πού βρίσκονται ακριβώς και για να ε, βρεθούν λύσεις. Και τέλος, για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Την υποστηρίζω. Αλλά για ποιο λόγο η Κομισιόν μιλά πάντοτε για την προστασία των καταναλωτών και όχι για την ενίσχυση των καταναλωτών. Γιατί υπάρχουν πλέον ε, ιστοσελίδες όπου μπορούν, μπορεί κανείς να ε, αξιολογεί ε, όλα τα προϊόντα που αγοράζει. Γιατί είναι και αυτό ένας, ε, ένα μέσο ε, για την προστασία των καταναλωτών. Και τέλος, ο Επίτροπος Έτιγκερ ε, έκανε την προηγούμενη εβδομάδα κάποια σχόλια που με ανησύχησαν γιατί ε, είπε ότι η Κομισιόν θέλει να προστατεύσει τους παίκτες στην, που βρίσκονται στην αγορά. Εμένα το ερώτημά μου είναι πώς μπορούν να προστατευθούν ε, οι ίσοι όροι ανταγωνισμού στην αγορά και όχι μόνο αυτούς που ήδη δραστηριοποιούνται στην αγορά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, είναι αστείο γιατί δεν ήξερα τι θα έλεγε ο συνάδελφος Τάλτον, αν και γνωρίζοντας ε, επί ποιο σημείο εργάζεται θα μπορούσα να το είχα φανταστεί. Θα απηχήσω βέβαια τα όσα είπε και εκείνο. Μιλήσατε αρχικά για επενδύσει. Ναι, είναι στρατηγική σημασία και λείπουν οι επενδύσει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ξέρουμε, για να μπορέσουμε να έχουμε ανάπτυξη και απασχόληση. Μιλήσατε για προγράμματα για τις επενδύσεις, αλλά για να έχουν αντίκτυπο οι επενδύσεις σε όλους τους τομείς των επιχειρήσεων θα πρέπει να γίνουν πιστευτές από όλο τον οργανωτικό μηχανισμό που υπάρχει από πίσω. Δηλαδή να πιστεύουμε στις αγορές πίσω από αυτά τα projects. Εδώ βρισκόμαστε στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και γι' αυτό και απηχώ ε, αυτό που είπε ο συνάδελφος Ντάλτον, ότι δηλαδή το θέμα των ε, μη δασμολογικών ε, φραγμών και εμποδίων είναι στρατηγική σημασία. Σα άκουσα που είπατε πριν από λίγο για startup, για τι νεοφυεί εταιρείε. γιατί μιλάμε συχνά για τι μεγάλε επιχειρήσει, αλλά ξεχνάμε τι ενδιάμεσε, δηλαδή τι μικρομεσαίε. Γιατί ακριβώ μέσω τη ανάπτυξη των μικρομεσαίων, ώστε μετά να φτάσουν σε ένα μεσαίο μέγεθο, όπου θα κρυθεί η δυνατότητα να γίνει και να υπάρξει αυτή η ανάπτυξη. Και γι' αυτό και σας θέτω πολύ συγκεκριμένο ερώτημα. Ποια μέσα, ποια εργαλεία, ποιες διατάξεις γιατί εγώ προέρχομαι από μια χώρα, τη Γαλλία, όπου συχνά μιλάμε για υπερβολική μεταγραφή των νομοθεσιών και πιστεύω πως αυτή τη στιγμή στη χώρα μου αλλά και στις άλλες χώρες αυτή η υπερβολική νομοθέτηση ε, είναι ένα δηλητήριο που δεν επιτρέπει να άρουμε τους δασμολογικούς φραγμούς. Αντίθετα προσθέτει και άλλος και πολύ συχνά με όλες τις καλές προθέσεις ε, και όχι φυσικά κατά των επιχειρήσεων. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι συγκεκριμένο με τους συναδέλφους σας. Ε, και ε, το σύνολο της Επιτροπής πώς θα μπορέσετε ακριβώς να αντιμετωπίσετε αυτό το τομέα και αυτό το πρόβλημα. Η Τζούλια Ρέιντα από τον πρώτο ε, γύρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Φυσικά έχετε πολύ σημαντικό ε, χαρτοφυλάκιο για αυτή την Επιτροπή και για την στρατηγική ψηφιακή ενιαίας αγοράς. Θα θέσω και πάλι το θέμα της ταχύτητας των μεταρρυθμίσεων όπως αυτές ε, προκύπτουν. Ε, μόλις ε, σήμερα ανεφέρθη ότι ένα από τα σημαντικά στοιχεία της στρατηγικής της Λισαβόνας, η μεταρρύθμιση του copyright, θα αναβληθεί για άλλη μια φορά και αυτή τη φορά για το Σεπτέμβριο. Οπότε Δεδομένου ότι ο πρόεδρος Γιούνκερ είχε ανακοινώσει πως η πρότασή του θα ερχόταν έξι μήνες μετά από την ανάληψη καθηκόντων, ενώ τώρα η, ε, βλέπουμε ότι η συμμόρφωση προς τις ε, προαναγγελίες είναι της τάξης του 4 Σκοπεύετε να κάνετε άλλη μια διαβούλευση ε, για το θέμα των συγγενικών δικαιωμάτων για τους εκδότες τύπου. Είπατε ότι η Επιτροπή στοχεύει στο να μην ευνοήσει μόνο ένα μοντέλο επιχειρηματικό, ε, έναντι κάποιων άλλων. Και αυτή η έκθεση της ενιαίας αγοράς επίσης λέει ότι δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν νέες υποχρεώσεις ε, ώστε να χρηματοδοτείτε ή να επιδοτείτε ένα συγκεκριμένο μοντέλο εις βάρος των υπολείπων. Και γι' αυτό θα ήθελα να γνωρίζω από την μια πλευρά, εσείς θα ασκήσετε την απαραίτητη ε, καθοδήγηση ώστε να αρχίσουμε γρήγορα να εργαζόμαστε πάνω σε όλα αυτά και έπειτα τα αποτελέσματα της έκθεσης ε, ε, θα ληφθούν υπόψη ώστε να μην υποβάλουμε προτάσεις που και πάλι θα καθιστούν δύσκολο για δύσκολο τον ανταγωνισμό στην ενιαία ψηφιακή αγορά για τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Τέλος, εδώ κάνουμε πολλή δουλειά για να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα ανθρώπων με ειδικέ ανάγκες, μιλάμε για την οδηγία ε, πρόσβασης κτλ. Και το να καθυστερήσει μεταρρύθμιση για τα copyright σημαίνει πάλι αναβολή της εφαρμογής της συνθήκης του Μαρακές που προβλέπει ότι οι άνθρωποι με ε, δυσκολίες όρασης ε, θα μπορούν να διαβάζουν ηλεκτρονικά βιβλία. Ε, υποτίθεται ότι αυτή η πρόταση είναι έτοιμη από το περασμένο Σεπτέμβριο και κάθεται σε κάποιο γραφείο της Κομισιόν. Θα εξασφαλίσετε ότι αυτή η πρόταση θα έρθει, θα κατατεθεί εδώ πριν το Σεπτέμβριο. Δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε και υπάρχει πλήρη στήριξη του Κοινοβουλίου για να προχωρήσει αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ μου αρέσουν τέτοιες συζητήσεις. Ε, είναι πολιτικής φύσης. Αντιλαμβάνομαι τις ανησυχίες σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω τις ερωτήσεις σας με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια, αλλά δεν γνωρίζω τις απαντήσεις πλήρως σε όλα τα ζητήματα που αναφέρατε, αλλά θα προσπαθήσω. Πρώτα απ' όλα για τη διαδικασία κοινοποίηση. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε την τρέχουσα υποχρέωση κοινοποίηση ε, στην οδηγία για τις υπηρεσίες. Οι νέες ή τροποποιημένες ε, απαιτήσει για τους πρώτους υπηρεσιών στα κράτη-μέλη είναι σημαντικό να κοινοποιούνται ώστε να είναι δυνατή η εισαγωγή αυτών των ε, μέτρων που μπορεί να επηρεάσουν την παροχή υπηρεσιών διασυνοριακά. Όσον αφορά τις πιο αποτελεσματικές διαδικασίες, ε, καλύπτουμε ε, ευρύ φάσμα απαιτήσεων ε, και δίνουμε και τη δυνατότητα στην Επιτροπή και στα κράτη-μέλη να εξετάζουν και να σχολιάζουν τα σχέδια εθνικών μέτρων, ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη λειτουργία της αγοράς υπηρεσιών. Στόχος μας λοιπόν είναι να αυξηθεί η διαφάνεια και να υπάρχει δυνατότητα αξιολόγηση της αναλογικότητας των νομιμέτρων. Η δεξιότητα, η, το θεματολόγιο για τις δεξιότητες, η ατζέντα δεξιοτήτων. Η Μαριάν Τάισαν ε, θα κάνει μια πρόταση για το θέμα αυτό του Skills Agenda μέσα σε λίγες εβδομάδες από τώρα. Εμείς ε, Προσπαθήσαμε να συνεργαστούμε. Ε, έχουμε συναντήθει πολλές φορές ε, για να συζητήσουμε και να καλύψουμε ολόκληρα το φάσμα των δεξιοτήτων. όπως για παράδειγμα δεξιότητες που απαιτούνται για την βελτίωση της παραγωγικότητας συγκεκριμένων βιομηχανιών, στη Χαλιβουργία για παράδειγμα. Όλοι συμφωνούν ε, για το βασικό ζήτημα. Αλλά ε, η Κομισιόν ε, δεν ξέρει τι να πει ότι μπορούμε να βελτιώσουμε, γιατί ξέρετε αυτή η πολιτική δεν είναι στα χέρια μας. Φυσικά μπορούμε να κοινοποιούμε, να κοινοποιούμε τις βέλτιστες πρακτικές της μίας χώρας σε μια άλλη ή να παρέχουμε συμβουλές στα κράτη-μέλη ε, να χρησιμοποιήσουν ως χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βελτιώσουν την ποιότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ε, παραδείγματι. Και ο ιδιωτικό τομέα παίζει σημαντικό ρόλο. Ε, Αυτό ο ιδιωτικό τομέα ορισμένε φορέ μπορεί να παρέχει πολύ πιο ευέλικτα την εκπαίδευση από ότι καθιερωμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Δεν λέω ότι θα αντικαταστηθούν οι σχολές από ιδιωτικές εταιρείε. Απλά μπορούν να παράσχουν επιπλέον βοήθεια για την επίλυση αυτού του ζητήματος. για αυτό το ευρύ θέμα θα μάθετε και θα ακούσετε και περισσότερα στο μέλλον. Να προσθέσω κάτι σε αυτό το σημαντικό θέμα της ατζέντα για τις δεξιότητε. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια τεράστια εισρωή ανθρώπων στην Ευρώπη και πρέπει να προσπαθήσουμε να του βοηθήσουμε να του εντάξουμε το ταχύτερο δυνατόν στις κοινωνίες μας ώστε και αυτοί να αρχίσουν να συμβάλλουν και να συμμετέχουν στι κοινωνίε μας. Από την αυσή τη ανταγωνιστικότητα και τη επένδυση, αυτοί οι άνθρωποι αποτελούν προσόν για τις χώρες μας, όχι μόνο βάρο, μπορούν να αποτελέσουν και προσόν για την Ήπειρό μας η οποία πιστεύει στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τώρα δέχεται ξαφνικά ε, πολλούς ανθρώπους αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτό το ανθρώπινο κεφάλαιο θα συνεχίσει να υπάρχει και στο μέλλον ε, και θα διατηρηθεί. Γι' αυτό το λόγο έχουμε μια νέα πρόκληση στην ατζέντα για τις δεξιότητες ε, όλο και περισσότερος κόσμος θα πρέπει να εκπαιδευτεί καλύτερα. Ε, για τη βελτίωση της νομοθεσίας, το Better Regulation, και τα ζητήματα των μη δασμολογικών φραγμών. Ε, η βελτίωση της νομοθεσίας το Better Regulation για πολλούς ε, σημαίνει σημαίνει ότι καταργούμε κάποιους κανονισμούς και έτσι μετράμε το, η βελτίωση ε, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ε, βελτίωση νομοθεσία σημαίνει και πολύ στενή συνεργασία με διάφορους τομεί ε, κατά την κατάρτιση νέων ε, κανονισμών. Για παράδειγμα, αν ο σκοπός μας ε, είναι να δημιουργήσουμε μια ενιαία αγορά, αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να αντικαταστήσουμε 28 κανονισμούς από έναν. Αυτό είναι ο καλύτερο τρόπος ε, αντιμετώπισης του διοικητικού άκθους αλλά φυσικά πρέπει η μία αυτή η νέα πρόταση να λαμβάνει υπόψη και τις διαφορετικές απόψεις. Ε, μπορεί να διαφωνήσετε με αυτό που θα πω, αλλά πρέπει να πω ότι η νέα μεθόδος εργασίας της Κομισιόν που διαφέρει από τη μεθόδο εργασίας προηγούμενης διότι έχουμε ομάδες έργων, project teams, αυτός ο νέος τρόπος εργασίας υποτίθεται θα βελτιώσει την ποιότητα των προτάσεων που θα παρουσιάζονται. Εγώ μαζί με τον κύριο Τίμερμανς ε, ε, ηγηθήκαμε ενός από, από τα βασικότερα προγράμματα της ενιαίας αγοράς που δεν θεωρείται πάντα θέμα της ενιαίας αγοράς βέβαια ε, πρόκειται για το πρόγραμμα της περικυκλικής οικονομίας ξέρετε, τα ζητήματα που εξετάστηκαν εκεί δεν, ήταν μόνο, δεν αφορούσαν μόνο το περιβάλλον, αλλά και την ενιαία αγορά. Οπότε πολλέ διαφορετικέ γενικέ διευθύνσει τη Κομισιόν συμμετείχαν. Και πρέπει να σα πω ότι το αποτέλεσμα ήταν πολύ καλύτερο από ότι η αρχική πρόταση. Οπότε έτσι βλέπω εγώ τη βελτίωση τη νομοθεσία, το Better Regulation. Ε, το ότι λαμβάνουμε υπόψη διαφορετικέ απόψει, αλλά όχι μόνο απόψει και διαφορετικέ οπτικές γωνίες. Δηλαδή η κυκλική οικονομία, ναι, έχουμε κάτι κυκλικό, κάτι που κυκλοφορεί, αλλά υπάρχει και η οικονομία, υπάρχει και η πτυχή της οικονομίας μέσα σε αυτό. Η μη δεσμολογική φραγμή τώρα Δεν σκέφτηκα κάτι για την πρόταση που λέτε εσεί, αλλά ούτω ή πρέπει να γίνει κάτι για, για του μη δασμολογικού φραγμού. Επειδή όπω όλοι εδώ ξέρετε, μία από τι προκλήσει που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι τα κράτη-μέλη δεν υλοποιούν ολόκληρη την νομοθεσία για την ενιαία αγορά. Και αυτό ακριβώ είναι ο λόγο που εμεί προτείναμε νέα εργαλεία. ώστε να επιτηρούμε ε, αυτά που κάνουν τα κράτη-μέλη αλλά και να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να ε, εφαρμόζουν τις νομοθεσίες αυτές. Ε, αυτή είναι μια από τις στρατηγικές της ενίας αγοράς. Οπότε εμείς ως Κομισιόν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα από ό,τι έχουμε κάνει στο παρελθόν αλλά υπολογίζω και στη δική σας υποστήριξη για το θέμα αυτό. Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προτεραιότητα σε αυτά τα ζητήματα υλοποίηση και εφαρμογή στην πολιτική ατζέντα. Δεν είναι κάτι καινούριο. Ε, μπορεί να μην είναι τόσο ενδιαφέρον διότι το έχουμε συζητήσει και ξαναζητήσει είναι παλιό θέμα αλλά είναι πολύ σημαντικό όπως είπα λοιπόν πρέπει να κάνουμε κάτι σε αυτό το μέτωπο οπωσδήποτε επίσης θέξατε το σημαντικό, το σημαντικό ζήτημα της ενδυνάμωσης των καταναλωτών αποτελεί αυτό το κομμάτι της κυκλικής ε, της οικονομίας και της σχετικής νοοτροπίας φυσικά Πρέπει να διασφαλίζουμε την προστασία των καταναλωτών. Αλλά πρέπει να παρέχουμε και κάποιο περιθώριο για επιλογές στους καταναλωτές. Η Ευρώπη είναι μια ήπειρος που επιτρέπει την εμφάνιση νέων ε, επιχειρηματικών μοντέλων. Είμαστε μια ήπειρος που έχει ορίσει ήδη τα μοντέλα και τις υπηρεσίες που μπορούν να παρέχονται στους καταναλωτές. Μας αρέσει ή όχι η συνεργατική οικονομία, για παράδειγμα, θα αρχίσει να αποκτά όλο και μεγαλύτερο ρόλο και εμείς θα πρέπει να βλέπουμε την Ευρώπη ως μια ήπειρο ασφαλή και ανοιχτή για νέες επιχειρηματικές προτάσεις. Γι' αυτό το λόγο τον Απρίλιο θα παρουσιάσουμε ένα έγγραφο, ε, τον Ιούνιο, συγγνώμη, ε, σε σχέση με τη συνεργατική οικονομία. Πώς εφαρμόζεται δηλαδή και η τρέχουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία στα νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Και εκεί σε Εντό αυτής τη κυκλική οικονομική και της συνεργατική οικονομίας εντάσσεται η ενδυνάμωση του καταναλωτή. Ε, ρωτήσετε και κάτι για τους μη δασμολογικούς φραγμού. Ελπίζω να κάλυψα έστω και μερικώ την ερώτησή σας. Yes. The copyright issue. Για το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων. Γνωρίζω ότι υπάρχουν δύο φάσεις που έχουν προγραμματιστεί. Ο εξυγχρονισμός του copyright πρώτα. Την προηγούμενη χρονιά προτείναμε μια μεταρρύθμιση της σχετικής νομοθεσίας. Και υποβάλαμε και μια νομοθετική πρόταση για την φορητότητα. το δεύτερο μεγάλο πακέτο μέτρων που πρόκειται να υποβάλουμε θα έρθει το καλοκαίρι. Δεν μπορώ να σας πω αν θα είναι Ιούνιος ή Ιούλιος, πάντως φέτος το καλοκαίρι θα γίνει. Και ο αντιπρόεδρος Άνσιπ δραστηριοποιείται ενεργά. Δεν έχουμε ε, κάποια εμπόδια Απλά θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι το πακέτο μέτρων που θα προτείνουμε θα είναι υψηλή ποιότητας. Και σας ευχαριστώ για την θετική σας στάση. Και κάτι τελευταίο που προέκυψε από τις προτάσεις για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Ο ρόλος της Επιτροπής σας θα είναι εξαιρετικά σημαντικός. στον τομέα αυτό. Γιατί είναι πάντοτε πολύ εύκολο να απορρίπτουμε προτάσεις που ενδεχομένως να αποδειχθούν δύσκολες ε, από κάποιες απόψεις και να χάνουμε τον βασικό στόχο που είναι η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. Εμείς δηλαδή θέλουμε να ε, συζητήσουμε με τους εμπλεκόμενους φορείς, με τα θεσμικά όργανα, αν η πρότασή μας έχει και ελαττώματα, ώστε σε δύο-τρία χρόνια να μπορέσουμε να έχουμε καταλήξει σε μια πολύ συγκεκριμένη ε, κατάληξη σε αυτό το θέμα. Για, τα, για τις ε, τρίτες χώρες και τη συμμετοχή τους ε, στο ΕΦΣΙ και την στρατηγική 2020 ε, είναι μια ερώτηση που την ξεχάσατε να την απαντήσετε. Ε, δεν ξέρω ποια είναι η επίσημη γραμμή για σήμερα. Δεν ξέρω τι μπορώ να σας πω επίσημα αυτή τη στιγμή. Ε, πάντως όλοι εδώ γνωρίζουν ότι σε κάθε περίπτωση τα κράτη-μέλη ε, τα μέλη, εν πάση περιπτώσει, οποιασδήποτε λέσχη κρατών, πάντοτε έχουν κατά προτεραιότητα πρόσβαση στα ωφέλη από ότι τα μη μέλη. Άνιτ Στέφανιτς και μετά ο Νίκολα Ντάντη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε για τις ε, σαφείς σας τοποθετήσεις σχετικά με την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Τρία θέματα θέλω να θέσω. Πρώτα απ' όλα είπατε ότι υπάρχουν 56 προγράμματα που έχουν εγκριθεί. Το ερώτημα μου είναι πόσα από αυτά αφορούν τον ε, ψηφιακό τομέα. Γιατί συμφωνούμε όλοι ότι η ψηφιακή ενιαία αγορά είναι προτεραιότητα, αλλά το ερώτημα είναι επίσης αν υποστηρίζονται ε, συγκεκριμένα έργα με βάση αυτή την προτεραιότητα. Και επίσης έχουμε μηχανισμούς μέσα για να διαμορφώσουμε στρατηγικές επενδύσεις για να υποστηριχθούν οι στρατηγικές μας προτεραιότητες στον τομέα ε, της ε, ψηφιακής τεχνολογίας. Δεύτερον, χάρηκα που είπατε ε, ότι υποστηρίζετε την απλούστευση του ΦΠΑ. Επίσης όμως θα ήθελα να σας ρωτήσω η Κομισιόν θα υποβάλει ε, πρόταση για την ενιαοποίηση της καταχώρησης ε, ΦΠΑ. Υποστηρίζεται κάποια τυποποίηση σε αυτό τον, ε, στον τομέα αυτό. Για τη χαλιβουργία. Είπατε ότι αντιμετωπίζει ισχυρές πιέσεις λόγω των εισαγωγών που βρίσκονται εισάγονται προϊόντα ε, κάτω του κόστους και νομίζω ότι χρειάζονται συντονισμένες προσπάθειες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Νίκολα Ντάντε. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Εσείς ε, περιγράψατε πολλά θέματα στο, που ανεμπίπτουν στο χαρτοφυλάκιό σας. Θα ήθελα εγώ να έχω την γνώμη σας για τα εξή τρία σημεία. Για το σχέδιο επενδύσεων είναι σημαντικό και ήδη δώσατε κάποια νούμερα που αρχίζουν να είναι σημαντικά. Θα χρειαζόταν κανονικά μεγαλύτερη ποσότητα, <clears throat> μεγαλύτερος όγκος πόρων, αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν. Ήταν ε, λίγα τα χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μα. αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε από ποιοτική άποψη. Αυτέ αυτές οι επενδύσεις που γίνονται είναι επενδύσεις με κάποιο κίνδυνο ή είναι επενδύσεις που ούτως ή άλλως θα τις είχαν κάνει οι ε, επιχειρήσεις γιατί ήταν ε, πόροι τους οποίους ε, θα μπορούσαν κάλλιστα να έχουν πάρει από την BAY, ε, την ΕΤΕΠ ή κάποια άλλη τράπεζα. Θέλω να γνωρίζω λοιπόν είναι κάποιες πιο επικίνδυνες επενδύσεις από τις πορείες μπορεί να έχουμε μια ανάπτυξη πραγματική μεγαλύτερη από ότι αν πηγαίναμε σε σίγουρες επενδύσεις. Δεύτερον, υπάρχουν κάποιοι κανόνες και κάποιες μελέτες της Επιτροπής που λένε ότι μπορούμε, τι μπορούμε να κάνουμε για να υπάρξει ανάκαμψη σε ορισμένου τομεί πράγματα αρκετά απλά. Και παραθέτω δύο. Πρώτο, πακέτο ε, εποπτείας της αγοράς και ε, made in. Και δεν το λέω εγώ ως καλός ε, μεσογειακός τύπος, αλλά το λένε οι μελέτες της Κομισιόν, που λένε μάλιστα ότι είναι πολύ καλά αυτά τα μέτρα. Ξέρω πως είναι εξάρτητα από την Κομισιόν, αλλά από το Συμβούλιο. Αλλά σας ρωτώ, η Κομισιόν τι κάνει για να διευκολύνει μια συμφωνία ανάμεσα στη θέση του Κοινοβουλίου και τη θέση του Συμβουλίου, τουλάχιστον για ορισμένου το Τελευταίο σημείο είναι εκείνο για την επέκταση των γεωγραφικών ενδείξεων. Το, δεν το λέει το Κοινοβούλιο, αν και το Κοινοβούλιο υπερψήφισε με 600 ψήφους υπέρ την πρόταση αυτή. Το λένε όμως και οι μελέτες της Κομισιόν ότι εδώ μπορούμε να έχουμε μικρές, όχι τελάστιες αυξήσεις του ΑΕΠ, αλλά μικρές αυξήσεις του ΑΕΠ. Υπάρχει συμφωνία στο Συμβούλιο, υπάρχει συμφωνία στο Ευρωκοινοβούλιο. Τι περιμένει η Κομισιόν για να υποβάλει νομοθετική πρόταση. Ευχαριστώ. Κυρία Βεργενή Ροζιέρ, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε που είστε εδώ. Εγώ θέλω να μιλήσω μόνο για το θέμα των ε, γεωγραφικών ενδείξεων. Ε, εδώ και έξι μήνες στο Κοινοβούλιο ε, γκρίναμε μια έκθεση της οποίας ήμουν μάλιστα εγώ εισηγήτρια με πολύ μεγάλη πλειοψηφία για την επέκταση των γεωγραφικών ενδείξεων. Το ίδιο ζήτησαν και η Επιτροπή Περιφερειών και η Οικονομική και η Κοινωνική. Μπορείτε να σηκώσετε λίγο το μικρόφωνο σας παρακαλώ γιατί δεν ακούγεστε πολύ καλά. Μάλιστα. Η Επιτροπή των Περιφερειών λοιπόν και η ΟΚΕ το ζήτησαν το ίδιο, αλλά η Κομισιόν στη μελέτη της του 2013 κατέληγε στη σκοπιμότητα ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για τις μη γεωργικές γεωγραφικές ενδείξεις και στην ανακοίνωσή σας ε, πριν από έξι μήνες είπατε ότι θέλατε να δώσετε συνέχεια σε αυτή τη διαβούλευση που τελείωσε στα τέλη του 2014 και που ήταν ευνοϊκή προς αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Είναι ένα θέμα για το οποίο πολύ συχνά με ρωτάνε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναμένουν αυτή την προστασία γιατί έχουν να αντιμετωπίσουν αθέμητο ανταγωνισμό από προϊόντα που κατασκευάζονται εκτός Ευρώπης που δεν έχουν καμιά σχέση με τα ευρωπαϊκά παραδοσιακά προϊόντα. Μέχρι στιγμής ε, η αναμονή ήταν, ε, ε, κάπου, ήταν με καλή θέληση αλλά τώρα αρχίζει να γίνεται ενόχληση πια. Δεν θα ήθελα λοιπόν να υποβαθμιστούν όλες αυτές οι επιχειρήσεις λόγω του χρόνου που μας παίρνει εμά για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες τους. Θέλω να ξέρω λοιπόν πότε θα έχουμε κοινό πλαίσιο λοιπόν για τις γεωγραφικές ενδείξεις για τα μη γεωργικά προϊόντα. Φανίστε Ρόι. Κύριε Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε. Είστε ο άνθρωπος του πολλαπλασιαστή. Με τα ταμείο αυτό πολλά πράγματα έχουν ήδη αλλάξει έστει ώστε να προωθηθούν ε, ιδιωτικό χρήμα στην οικονομία. Θέλω να μιλήσω για, το, για τις startups και τις scale-ups. Έχουμε πολλές ε, νεοφύης εταιρείε σε διάφορους τομείς, αλλά το θέμα είναι ότι ανάμεσα στα 10 και στα 100 εκατομμύρια δεν μπορείς να συγκρίνεις με τις ΙΠΑ. Είμαστε πολύ πίσω. Και αυτό εδώ λέτε 75 δις πάνε από τα κράτη-μέλη, από, τα, από τους κόμβους, τα hubs και κάθε εβδομάδα ανακοινώνεται τι γίνεται. Πώς προχωράνε αυτά τα πράγματα. Έχετε πραγματικά ανοιχτή σύνδεση με τις startups και τις scale-ups. Και η τελευταία μου ερώτηση είναι το εξή. Μπορούμε να κάνουμε πολλά μεγάλα βήματα για νέα προϊόντα, με βιολογικά προϊόντα, από τη στιγμή που όμως δεν έχουμε μια τέτοια ενιαία αγορά για το τι είναι απόβλητο και τι δεν είναι απόβλητο επικρατεί σύγχυση και χάνουμε πολλές ευκαιρίες. Εγώ λοιπόν υποστηρίζω αυτό το συνδυασμό στο χαρτοφυλάκιό σας. Does Άλλος θέλει το λόγο. Να προσθέσω κι εγώ δύο παρατηρήσεις. Καταρχήν για το διαβατήριο των υπηρεσιών. Εμένα μου αρέσει αυτή η ιδέα να υπάρχει ένα διαβατήριο για τις υπηρεσίες που σημαίνει δηλαδή ότι χρειάζεται μόνο απόδειξη ότι μπορείς να βρίσκεσαι, σε, ότι είσαι σε ένα κράτος μέλος και μπορείς να το περάσεις και στα υπόλοιπα 28. Όμως γνωρίζουμε ότι αυτός ο τομέας αντιπροσωπεύει πολλές μικρομεσαίες που λένε ότι δεν το θέλουν γιατί πιστεύουν ότι θα καταλήξει σε εξαιρετικά περίπλοκο ε, διχασμό ανατομέα στις υπηρεσίες και ότι θα κολλήσουμε στις διαπραγματεύσεις. Υπάρχει λοιπόν πολύ διαφορετική άποψη για το τι σημαίνει το διαβατήριο των υπηρεσιών για μερικού από εμά και τι θέλουν εκείνοι. Άρα λοιπόν η ερώτησή μου είναι μπορούμε περισσότερο χρόνο να περάσουμε με τους άμεσα ενδιαφερόμενους γιατί ε, ε, θα πρέπει να έχουμε μια επαφή με τους πραγματικούς παρόμοιθευτές των ε, παρόχους των υπηρεσιών. Να υπάρχει συνεργασία, να υπάρχει διασυνοριακή ενημέρωση και τα πόρταλ που φτιάχτηκαν ή μάλλον θα φτιαχτούν σύμφωνα με την ε, οδηγία των υπηρεσιών να λειτουργούν ώστε να μπορούν πράγματι οι πάροχοι των υπηρεσιών να έχουν τις πληροφορίες στη θέση τους. Γιατί δεν το υποστηρίζουν λοιπόν Και έπειτα, για την ατζέντα της καλύτερης νομοθεσίας. Άκουσα με χαρά ότι υπάρχει ελπίδα ότι περισσότερη έλλειψη γραφειοκρατίας θα προέλθει από την καλύτερη διαβούλευση από κάτω προς τα πάνω μέσα του της πλατφόρμας Refit. Μπήκα και βρίδα το Refit και αυτή την εκστρατεία γιατί θέλω να ενθαρρύνω τον κόσμο αν έχουν δει που κάπου υπερβολική γραφειοκρατία να το αναφέρουν. Αλλά είναι τόσο περίπλοκο αυτό το site που πρέπει κανείς να βάλει EC, Europe κτλ. Δημοκρατικές αλλαγές ε, ε, κτλ. Εν πάση περιπτώσει, για να βρεις και μόνο το site πρέπει να είσαι ταχυδακτυλουργός. Ε, άρα λοιπόν το βρίσκω πολύ δύσκολο να πω αυτό όλο το όνομα του site σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, ας πούμε, να κάνω διαφήμιση. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η σύντομη ε, μια σύντομη, ένα σύντομο site, όνομα μάλλον για το site, να λέει «Cut red tape». Ε, κόψτε τη γραφειοκρατία, μειώστε τη γραφειοκρατία. Κάτι πιο σύντομο και πιο εύκολο. Ναι, πολύ καλή ιδέα. Ευχαριστώ πολύ. Για τα ψηφιακά προγράμματα, γύρω στο 10% ή λιγότερο το των project που έχουν χρηματοδοτηθεί αφορούν το ψηφιακό τομέα. Όταν ξεκίνησε το ΕΦΣΥ, εγώ είχα φανταστεί πως ήταν περισσότερο το τμήμα αυτό, ότι δηλαδή οι ψηφιακές επενδύσεις ήταν περισσότερες, αλλά μέχρι στιγμής δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω στα προετοιμαζόμενα προγράμματα, εάν υπάρχουν και άλλα ψηφιακά, αλλά πάντως μέχρι στιγμής αυτό είναι το νούμερο. Τα περισσότερα προγράμματα του ΕΦΣΙ έχουν να κάνουν με την ενέργεια, με νέες ενέργειες, με φυή πλέγματα κτλ. κτλ. Ίσως να χρειάζεται κάποια όθηση στο ψηφιακό site, αν και δεν είναι η Κομισιόν αυτή που επιλέγει τα project. Είναι ένα ταμείο που κινείται με βάση τη ζήτηση. Θα πρέπει να υπάρχει δηλαδή αντίστοιχη ζήτηση από πλευρά των επενδυτών. Ε, ίσως όμως θα έπρεπε εμείς να το προωθήσουμε με κάποιο τρόπο. Μια τώρα ευκαιρία για να προωθηθούν οι ψηφιακές επενδύσεις, ιδιαίτερα σε ορισμένες χώρες της συνοχής, είναι να χρησιμοποιηθούν τα διαστατικά ταμεία μαζί με το ΕΦΣΥ. Και εκεί θα μπορούσα να φανταστώ κάποιες ε, βασικές και απαραίτητες επενδύσεις υποδομών που θα μπορούσαν όντως να χρηματοδοτηθούν. Και θα ε, σήμαινε ότι και Εκεί θα συμμετείχαν και ιδιώτες επενδυτές. Ε, δυστυχώς δεν μπορώ να σας απαντήσω για το ε, δεύτερο σας ερώτημα, αλλά θα επανέλθω. Τώρα, χαλιβουργία. Πολύ περίπλοκο θέμα και γι' αυτό μάλιστα την Τετάρτη θα δημοσιεύσουμε μια ανακοίνωση γι' αυτό το θέμα, όπου θα παραθέσουμε μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει ισότιμο πεδίο για όλους ή θα, εν περιπτώσει, θα λάβουμε υπόψη τις αρνητικές επιπτώσεις της υπερπαραγωγής σε ορισμένες χώρες, ιδιαίτερα στην Κίνα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να επαγρυπνούμε για αυτό το θέμα, διότι οι τάσεις είναι εξαιρετικά έντονες. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα με ένα-δύο μέτρα. Θα πρέπει να έχουμε μια ολόκληρη παλέτα ε, μέτρων και μέσων. θα πρέπει να βοηθήσουμε και την ίδιο το κλάδο να επενδύσει στο μέλλον, ώστε να είναι πιο παραγωγικό. Θα επανέλθουμε σε αυτό, όπως σας είπα, την Τετάρτη. Επενδύσεις και εύση και κατά πόσο έχει δημιουργήσει προσθεθέμενη αξία. Αυτό είναι θέμα κλειδί. Γιατί όσοι έχουν συμμετέχει σε, αυτή τις, σε αυτές τις εργασίες ε, θεωρούν ότι είναι η προστιθέμενη αξία που είναι βασική. Η ΕΤΕΠ χρηματοδοτεί 70 δις ετησίως και το ΕΦΣΙ θα έπρεπε να έρθει να συμπληρώσει όλα αυτά και να εστιάσει σε διάφορους τομείς που να είναι οικονομικά βιώσιμοι, πιο σίγουροι αλλά και πιο επικίνδυνοι από ό,τι μπορεί να αναλάβει από μόνο στο ιδιωτικό τομέα. Έχω συζητήσει το θέμα μια-δυο φορές με τον ε, Διευθυντή Μόλτερν που είναι ο Διευθυντής της Επιτροπής Επενδύσεων του ΕΦΣΗ. και γνωρίζει πραγματικά ότι ισχύει αυτό και ότι για κάθε project που επιλέγουν φροντίζουν ώστε να είναι αρκετά καλό αλλά δεν έχει πλήρη χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα. Και αυτό είναι σημαντικό και από μια άλλη άποψη, διότι δεν θέλουμε να έρθουμε, μπούμε σε ανταγωνισμό με τον ιδιωτικό τομέα. Ο ιδιωτικό τομέα κάνει τη δουλειά του και του ενθαρρύνουμε. Αλλά υπάρχουν πάντα επενδύσει που είναι λίγο πιο ε, ή χρειάζονται δημόσια εγγύηση. Να σας δώσω ένα ενδιαφέρον ε, παράδειγμα. Ε, τι μπορούμε να κάνουμε. Στη Δανία έχουμε φτιάξει ένα, έχει φτιαχτεί ένα ταμείο το οποίο χρηματοδοτεί επενδύσεις ε, για την ανανεώσιμη πηγές ενέργειας στη Βόρεια Ευρώπη. Είναι ένα τα κονδύλι Η διαφορά με το ΕΦΣΥ είναι ότι βάζει τα χρήματα σε ένα χαμηλότερο θέμα, ε, σημείο και αυτό προσελκύει τα, τα συνταξιδοτικά ταμεία. Είναι η πρώτη φορά που ακούω στην Ένωση να γίνεται κάτι τέτοιο. Δηλαδή τα συνταξιδοτικά ταμεία να μπορούν να χρηματοδοτήσουν μικρότερα προγράμματα. Και εδώ προσθέτει ε, αξία το ΕΦΣΥ, χωρίς να ε, ε, χωρίς τα χρήματα του ΕΦΣΥ ποτέ τα συνταξιδοτικά ταμεία δεν θα ρισκάριζαν να μπουν σε τέτοια προγράμματα. Και τα όσα λέω μπορείτε φυσικά να τα παραθέσετε και να τα αναφέρετε και να τα διαδώσετε. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τη χρηματοδότηση από το ΕΦΣΥ, μπορείτε εύκολα να τα βρείτε στο site του ΕΦΣΥ και επανελειμμένα έχω επισκεφτεί εδώ το Κοινοβούλιο ως ομιλητή σε διάφορα ε, ε, που σε διάφορες εκδηλώσεις ώστε να μπορέσουμε να διαδώσουμε τις καλές πρακτικές ολόκληρη την Ευρώπη. για τις γεωγραφικές ενδείξεις αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τίποτα. Εγώ Μιλάω για γεωγραφικές ενδείξεις μόνο όταν συνομιλώ με τους Αμερικανούς για το TTIP. Και πάντα λέω ότι είναι μέρος της πρότασής μας, αλλά είναι αυτό εδώ που με ρωτήσατε τελείως διαφορετικό πράγμα. Μπορώ να σας στείλω τις απαντήσεις λοιπόν αργότερα, αν ε, μου το επιτρέπετε. Startups και scale-ups. Jonathan Hill, um, uh, uh, sorry, Carlos Moedas, Jonathan Hill will do a concrete proposal on uh, venture capital. Θα κάνουμε νέε προτάσει για το venture capital και τα διορθωτικά ταμεία, τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου δηλαδή και τα διορθωτικά ταμεία για να συλλέξουμε νέου πόρου, ώστε το μέγεθο του ταμείου να πλησιάζει τα 500 εκατομμύρια ευρώ τα μισά από τα οποία θα προερχόνται από το δημόσιο τομέα και τα υπόλοιπα από τον ιδιωτικό τομέα. Όλα αυτά για τι νεοφύης και τι επεκτενόμενες επιχειρήσει. Αυτή είναι μια από τι προτάσει που θα προκύψει, αν θυμάμαι καλά, μέχρι τι καλοκαιρινέ διακοπέ. Σκοπός λοιπόν ε, να δημιουργήσουμε ένα ευρύ ευρωπαϊκό ταμείο για επενδύσεις ε, ευρωπαϊκές και ενθάρρυνση ε, για μεγέθυνση των κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου των venture capital στην Ευρώπη σε μέγεθος που να φτάνουν τα αμερικάνικα τα οποία είναι πολύ υψηλότερα. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε αυτή τη μέθοδο και το εύση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τέτοια κλίμακα στόχων ε, και μπορεί να το πραγματοποιήσει και μέσω διαφορετικών ταμείων ή από μόνο του. Αυτό το μήνυμα λοιπόν πρέπει να το διαβιβάσετε στους κύκλους ε, των ε, ανθρώπων που ασχολούνται με κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου, με venture capitals. Τώρα το διαβατήριο για τις υπηρεσίες θα ξεκινήσουμε μια δημόσια διαβούλευση και ευχαριστούμε πάρα πολύ που αναφέρατε αυτές τις επικρίσεις γιατί θέλουμε να έχουμε τα σχόλια όσων πρόκειται να υποφεληθούν από αυτό το διαβατήριο για τις υπηρεσίες για να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Είμαστε πεπισμένοι ότι θα μπορούσαμε να το φτιάξουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθήσουμε ειδικότερα τους μικρού και μεσαίου μεγέθους παρόχους ε, υπηρεσιών στις διασυνοριακές τους συναλλαγές. Αλλά αν υπάρχουν ανησυχίες θέλουμε να τις ακούσουμε. Γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία ε, θα την ξεκινήσουμε μάλλον μέσω μιας δημόσιας διαβούλευσης. Ναι, έχουμε κάποια στοιχεία, υπάρχουν κάποιες προτάσεις, απλά εμείς θα εξηγήσουμε ουσιαστικά ε, ε, τι είχαμε εμείς στο νου μας, θα συλλέξουμε πληροφορίες και θα δούμε πού μπορούμε να προχωρήσουμε. Ελπίζουμε να βρούμε μια πολύ απλή μέθοδο που να βοηθήσει ουσιαστικά την επίτευξη των στόχων μέσω αυτής της συλλογής δεδομένων και στοιχείων από όλους. Ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει να βρούμε ένα καλύτερο όνομα για το cut red tape, έτσι πιο πιασάρικο. Γιατί αλλιώς θα φτύει ε, από την Κομισιόν και δεν νομίζω ότι αυτό είναι ο σκοπό σα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Επίτροπε που ήρθατε εδώ. Δεν ξέρω τώρα αν το γνωρίζουν τα μέλη. Όλα τα σχόλια από τις συζητήσεις του διαρθρωμένου διαλόγου Όλα αυτά τα στοιχεία συγκεντρώνονται στις συζητήσεις μεταξύ της διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών και των Επιτρόπων για την εκπόνηση του προγράμματος εργασιών. Οπότε το επόμενο φθινόπωρο όταν θα ξανασυναντηθούμε ε, σε μικροομάδες μεταξύ ε, ε, της διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών και ε, της ομάδας των επιτρόπων όλες οι ερωτήσεις που κάνατε εδώ σήμερα, που κάνετε εδώ γενικά λαμβάνονται υπόψη και μελτά καταλήγουμε σε κάποια συμπεράσματα βάσει των οποίων διαμορφώνεται το πρόγραμμα εργασιών για το επόμενο έτος. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικά τα σχόλιά σας. Ε, ευχαριστούμε που βρεθήκατε μαζί, μαζί μας. Um, now I will go to the... Λοιπόν, να περάσουμε στι ανακοινώσει του Προέδρου που συνήθω γίνεται στην αρχή τη συνάντηση, αλλά ήταν εδώ Επίτροπο. Λοιπόν, τρεις κλασικές ανακοινώσει. Υπενθύμηση, έχουμε, μεταδίδεται η συνάντηση live, η εφαρμογή meeting είναι διαθέσιμη για όλα τα μέλη, τους βοηθούς και τα μέλη του προσωπικού και η νέα ε, έκδοση του ενημερωτικού δελτίου, του newsletter έχει κυκλοφορήσει. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι ενημέρωση για τους τριμερείς διαλόγους αυτών που είχαμε για την προσβασιμότητα στις ιστοσελίδες των δημοσίων οργανισμών. Αλλά ο εισηγητής δεν βρίσκεται εδώ. Οπότε ας προχωρήσουμε και θα επανέλθουμε σε αυτό αργότερα. Ε, θα έρθει η εισηγήτρια. Όχι. Να δούμε πως βρούμε λίγο χρόνο αύριο για να το συζητήσουμε με την εισηγήτρια. Um, and then an on the Και μετά ενημέρωση για τον τριμερή διάλογο για τις ιατροτεχνολογικές συσκευέ και τις διαγνωστικές συσκευέ in vitro. Και θα γίνει μια ανακοίνωση εκ μέρους του Αντρέα Βάπ. Ανοίξτε την υπομονή, θα σας διαβάσω τα όσα έχει ετοιμάσει ο κ. Αντρέα Βάπ για σας. Ζητά συγγνώμη γιατί δεν μπόρεσα να βρεθεί εδώ σήμερα, αλλά προετοίμασα αυτό το εγγραφό το οποίο λέει τα εξή. Η ο έκτος τριμερής διάλογος ε, για τις ιατρικές συσκευές και τις τεχνολογικές συσκευές ε, in vitro έλαβε χώρα 17 Φεβρουαρίου του 2016. Πρόκειται για τον πρώτο υπό Ολλανδική Προεδρία. Όλες οι πλευρές αναμένουν να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις ε, στην τρέχουσα Προεδρία. Σχεδόν όλα τα κεφάλαια και τα παραρτήματα των δύο έχουν ανοιχτεί για διαπραγματεύσεις και οι συζητήσεις συνεχίστηκαν για πολλά σημαντικά ζητήματα. Το βασικό στοιχείο του έκτου τριμερούς διαλόγου από πλευράς ΙΜΚΟ ήταν η συζήτηση περί εξέτασης και πιο συγκεκριμένα το πεδίο εφαρμογής. Όσον αφορά το κεφάλαιο 5, εξέταση του ιατρικών συσκευών υψηλού κινδύνου, για το DS, δεν γνωρίζουμε λίτρια περί πρόκειται και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν ε, πετύχει συμβιβαστικό ε, κείμενο. Κατά τον τρίτο διάλογο, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε μια κοινή θέση για το πεδίο εφαρμογή και συμφώνησε έτσι να ε, αφήσει στην άκρη την τροπολογία για τους κοινοποιημένους οργανισμούς. Στην Κορεπέρ 26 Ιανουαρίου περιορίστηκε κάπως το πεδίο εφαρμογή ε, που πρότεινε το Κοινοβούλιο και τα κριτηρία βάση των οποίων η ομάδα εμπρογνωμόνων θα μπορούσε να επιλέξει την εφαρμογή της διαδικασίας. Επίσης ε, διαγράφηκε η διαταξή περί κατεξοδότηση πράξης που θα επέτρεπε στην Κομισιόν να αλλάξει το πεδίο εφαρμογή στο μέλλον. Το πεδίο εφαρμογή το Συμβούλιο αποδέχτηκε ευρύτερο πεδίο εφαρμογή όπως και ενεργές ε, συσκευές κλάσης 2Β, κλάσης 2Β. Αυτό καλύπτει και τις αντλήσεις ινσουλίνης. Αλλά φέρεσαν συσκευές που έχουν ε, κατασκευαστεί ε, χρησιμοποιώντας ιστούς ή κύτταρα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε να δεχθεί το προτινόμενο πεδίο εφαρμογή με μια διευκρίνηση στο κείμενο ώστε να διασφαλίζεται ότι όλες ε, οι συσκευές κλάσεις 3 και 2 θα καλύπτονται. Η κατεξουσιοδότηση πράξης τώρα για την επέκταση του εύρους εφαρμογής. Το Συμβούλιο διέγραψε αυτή τη διάταξη από την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν θέχθηκε να τροποποιηθεί κατά κανένα λόγο τρόπο το, εύρος, το επειδή εφαρμογής της διαδικασίας. Σε περίπτωση που κυκλοφορήσει μια νέα συσκευή που θα πρέπει να εξεταστεί πιο λεπτομερώς ε, λέει το Κοινοβούλιο ότι πρέπει να αναφέρει να περιγράφει αυτός ο τρόπος εξέτασης ε, και η όλη διαδικασία. Θα το εξετάσει το Κοινοβούλιο και θα επανέλθει γι' αυτό τώρα για τα τέλη η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν ότι οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να καταβάλουν τέλη για την κάλυψη των κόστους ε, επιπλέον κλινικών εξετάσεων. Η θέση του Συμβουλίου είναι ότι τα τέλη θα πρέπει να καταβάλλονται και να είναι χαμηλότερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε οι επιχειρήσεις να πληρώνουν το πολύ 50, το 50% του τέλους και το υπόλοιπο το καλύπτει κομισιόν. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, θα υπάρχει περαιτέρω έκπτωση από το 50% που πρέπει να καταβάλουν. Δεν έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής καμία συμφωνία η Κομισιόν εξέφρασε τις επιφυλάξεις της προς τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διότι συνεπαγόνται οι οικονομικές επιπτώσεις για την Κομισιόν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συζητήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάποιο δυνατό πιθανό συμβιβασμό. Η θέση του Συμβουλίου είναι ότι κάποιος πρέπει να πληρώσει τη διαδικασία και στην φάση αυτός θα είναι οι εταιρείε. Η θέση που ακολουθήθηκε είναι ότι όλες οι συσκευές θα πρέπει να αναφέρονται στην Κομισιόν η οποία θα αποφασίζει εντός 15 μερού βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων κατά πώ θα τις παραπέμψει στην ομάδα εμπειρογνώμων για περαιτέρω εξέταση. Το Συμβούλιο πρότεινε όλες, ε, όλα τα μηχανήματα, όλες οι συσκευές να παραπέμπονται απευθείας στην ομάδα εμπειρογνωμόνων με περιθώριο 21 ημερών για να αποφασίσει κατά πόσο θα εκδώσει η γνωμοδότηση. Επίσης το Συμβούλιο έχει κάνει πιο περιοριστικά τα κριτήρια επιπλέον εξέταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να δεχθεί τα πιο αυστηρά κριτήρια ενώ Συζητείται ακόμα η πρόταση του κ. Φάρελ στην ε, ομάδα εμπειρογνωμόνων και το Κοινοβούλιο προσπάθησε να απαντήσει την ερώτηση για το τι συμβαίνει όταν η ομάδα εμπειρογνωμόνων δεν εκδώσει ε, γνωμοδότηση εντός των 16 ημερών που έχει στη διάθεσή του. Και το τελευταίο έβριμα ε, είναι εξέταση για κλάση 4D διαδικασία που δεν προβλέπεται στην πρόταση του Συμβουλίου, διότι το Συμβούλιο θεωρεί ότι οι συσκευές υψηλότερου κινδύνου ήδη καλύπτονται από την τρέχουσα διάταξη. Αυτά υπάρχουν στο αρθρό 40, όπου όλες, ε, όλα τα μηχανήματα κλάσης D, ακόμη και χωρίς τεχνικές προδιαγραφές, θα πρέπει να υπόκειται στην εξέταση ενός Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Αναφοράς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εξετάσει την υπόθεση περαιτέρω μαζί με την Κομισιόν ε, για να δει κατά πόσο πράγματι η κλάση D χωρίς ε, προδιαγραφές ε, καλύπτεται έτσι όπως εξηγείται από το Συμβούλιο. Αυτά έστειλε ο Ανδρέας Φάβε. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστώ. Για να συνοψίσω, νομίζω ότι πολλοί έχουμε ανταλλάξει email και πληροφορίες γενικότερα για αυτήν την ε, οδηγία και ευχαριστούμε τον Ανδρέας που συνέταξε αυτό το έγγραφο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ιδίω ε, τι συμβαίνει με τις υπάρχουσες συσκευές. Στέντ, καρδιολογικά για παράδειγμα. Τι θα γίνει με αυτές, θα πρέπει να ξαναπεράσουν από μια διαδικασία έγκρισης, αδειοδότησης. Μήπως αυτό θα σημάνει ότι θα υπάρξουν καθυστερήσεις, ε, για να μπορούν οι καταναλωτές να αποκτήσουν κάποια από, αυτή, από αυτές τις συσκευές. Και ξέρω ότι ο Ανδρέας ενδιαφέρεται πολύ ώστε η οδηγία αυτή να μην δημιουργήσει προβλήματα κατά την εφαρμογή της. Θα πρέπει δηλαδή να εξασφαλίσουμε να καταλήξουμε και να τονίζεται η θέση της Επιτροπής ΙΜΚΟ η οποία είναι πάντοτε ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των καταναλωτών σε αυτού του είδους τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ακόμα και στη διαδικασία της μετάβασης. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η γνωμοδότηση για την ε, επίτευξη μιας νέας συμφωνίας για τους ε, καταναλωτές ενέργειας. Κάγια Κάλλας εισηγήτρια, 72 τροποποιήσεις, τροπολογίες έχουν υποβληθεί, 8 συμβιβαστικές τροπολογίες, αύριο θα γίνει ψηφοφορία και δίνω το λόγο στην Κάγια Κάλλας για να μας παρουσιάσει τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε 8 όπως είπατε συμβιβαστικές τροπολογίες, 2 εξ αυτών είναι νέοι συμβιβασμοί για να δοθεί ιδιαίτερη σημασία σε δύο σημαντικά θέματα που επισημάνθηκαν από τους συναδέλφους. Πρώτον, ότι ε, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ε, καμπάνιες για την συλλογική μετάβαση και η σημασία ε, των κανόνων ε, σχετικά με τους αθέμητους, τις αθέμητες πρακτικές ανταγωνισμού. Οι συμβιβασμοί επίσης αφορούν ε, την διαφάνεια και την ε, διάρθρωση των ε, τιμών. Ένα ζήτημα που μας ενδιαφέρει πολύ είναι ότι όταν οι καταναλωτές θέλουν δεν ωφελούνται ιδιαίτερα από τις διακυμάνσεις της κατανάλωσης τους γιατί υπάρχουν ανελαστικά κόστη που σχετίζονται με τη συντήρηση των δικτύων κτλ. Γι' αυτό άλλωστε ο κανονισμός για τις τιμές στην ουσία αυξάνει τις τιμές των, ε, της ενέργειας και γι' αυτό και καλούμε για την κατάργησή του την σταδιακή ε, και την ε, εξέταση της πιθανότητας να δημιουργηθούν νέοι μηχανισμοί και μέσα. Σε τελική ανάλυση όμως, ε, αν αποκτήσουμε μια αγορά που θα λειτουργεί στη βάση της αρχής ανταγωνιστικότητας, θα μειωθούν και οι τιμές για τους καταναλωτές. Επίσης, ε, θα πρέπει να υπάρξει και να καταρτιστεί μια φιλόδοξη πολιτική για την ενεργειακή αποδοτικότητα με ανακαινήσεις κτηρίων αλλά και με την δημιουργία ψηφιακών εργαλείων κάτι που επίσης θα μειώσει τις τιμές για τους τελικούς καταναλωτές. Συνολικά η ανακοίνωση της Κομισιόν είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο της κατανάλωσής τους οι καταναλωτές. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι θα πρέπει να γίνουν και ε, ενεργοί καταναλωτές, αλλά θα πρέπει τουλάχιστον να έχουν όλοι οι πολίτες στη διάθεσή τους τα εργαλεία εκείνα για να μπορούν να διαχειρίζονται την ε, κατανάλωσή τους όσον αφορά την ενέργεια. Περιμένω τα σχόλιά σας. Αντώνιο Λόπες είναι ο σκιώδης του ΕΛΚ, αλλά δεν βρίσκεται εδώ. αλλά δεν είναι εδώ, στην αίθουσα, όπως είπα. Μποζάν Μπελτζιάνα, σκιώδης των σοσιαλιστών, επίσης δεν είναι εδώ. Τεράστιο το ενδιαφέρον για το τι συμβαίνει στους λογαριασμούς των καταναλωτών και το τι πληρώνουν οι άνθρωποι. Εν πάση περιπτώσει. Ντάλιν, εσύ εκ μέρους του ECR μάλλον, έτσι. Ναι, ο κύριος Πρέτσελ είναι ο σκιώδης μας, προς το παρόν τουλάχιστον. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μπορούμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Κάλλας για το έργο της. Εμείς υποστηρίζουμε όλους τις συμβαστικές πρωτολογίες, ιδίως αυτές που αφορούν τη διαφάνεια και την ανταγωνιστικότητα και νομίζουμε ότι ένα από τα βασικά θέματα είναι ότι χρειαζόμαστε πλατφόρμες που θα επιτρέπουν στους καταναλωτές να κάνουν τη μετάβαση. Γιατί πολλοί καταναλωτές δεν κάνουν τη μετάβαση, γιατί δεν καταλαβαίνουν τι, ποιες είναι οι δυνατότητες που έχουν, τι, ποιες ε, επιλογές διατίθενται, άρα χρειάζονται εργαλεία για να μπορούν να συγκρίνουν και να κατανοούν το τι ακριβώς διατίθεται στην αγορά κάτι που θα τους δώσει και τη δυνατότητα να κάνουν τη μετάβαση. Ε, είχαμε κάποιες ε, διαφωνίες όσον αφορά την ενεργειακή ένδυα και την σχετική ορολογία. Ε, σε κάθε περίπτωση σε αυτό που συμφωνούμε είναι ότι ο ανταγωνισμός θα μειώσει τις τιμές και φαίνεται ότι στα, -μέλη, στα περισσότερα κράτη-μέλη δεν λειτουργεί παρκώς ο ανταγωνισμός. Ε, τέλος, λόγω της περιβαλλοντικής νομοθεσίας έχουμε καταλήξει να πληττόμαστε από το πρόβλημα της ε, ενεργειακής ε, φτώχειας και ε, διότι έχουν αυξηθεί, έχει αυξηθεί το κόστος της ενέργειας που πολύ συχνά όμως μετακυλίεται στους πιο ε, ευάλωτους καταναλωτές. Αυτά όσον αφορά την περιβαλλοντική νομοθεσία. Εν πάση περιπτώσει εμείς όπως είπα στηρίζουμε τις συμβαστικές τροπολογίες που υποβλήθηκαν και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με την εισηγήτρια. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο για αυτό το θέμα. Μπορούμε να περιμένουμε πάρα πολύ λίγο για να έρθει ο Αντώνιο, που είναι εσκιώδης εισηγητής εκ μέρους του ΕΛΚ. I'm so sorry. Is it, are you, are you yeah, yeah, yeah, yeah. Okay. Thank you very much. Thank you. Uh... Η κυρία Μπόζαν. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την συμβολή τους. Χαίρομαι που τα, οι περισσότερες ε, τροπολογίες προέρχονται από τους σοσιαλιστές. Πρέπει να πω ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τις ε, συμβαστικές τροπολογίες όσον αφορά τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές, γιατί όπως γνωρίζετε οι καταναλωτές πολύ συχνά γίνονται ε, θύματα ε, αθέμητων εμπορικών πρακτικών, ιδίως όσον αφορά τις ε, πωλήσει από πόρτα σε πόρτα. Γι' αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι καταναλωτές και να να τους δοθούν περισσότερες δυνατότητες επιλογής στην αγορά. Ε, οι σοσιαλιστές, όπως είπαμε και στην ε, συνάντηση των σκιωδών, θα υποστηρίξουν όλες τις τροπολογίες, εκτός από την τροπολογία 2. Γιατί οι ευάλωτοι καταναλωτές θεωρούμε ότι θα πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο και όχι να αφαιθούν στην τύχη της αγοράς. Είμαστε πάρα πολύ αυστηροί σε αυτό το θέμα και εμείς δεν μπορούμε να αποδεχτούμε τη συγκεκριμένη διατύπωση. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που πρόσθεσαν στοιχεία στην έκθεση, για παράδειγμα την τροπολογία της Λίζα για τα μονοπόλια ή άλλες τροπολογίες για τα τέλη μετάβασης. Σε κάθε περίπτωση οι θα πρέπει να, ε, η μετάβαση θα πρέπει να γίνεται με διαφάνεια, χωρίς να ε, υπάρχουν κρυμμένα τέλη ή κρυμμένες χρεώσεις, ιδίως από εκείνους που απολαμβάνουν κυρίαρχη θέση στην αγορά. Ευχαριστώ. Αντώνια. Αντώνιο. Εκ μέρους του ΕΛΚ, θέλεις να πάρεις το λόγο. Έχει γίνει ήδη ένας ε, γύρος τοποθετήσεων. Αλλά είμαστε στη διάθεσή σου να σε ακούσουμε. Παρακαλώ. Ήταν ακριβώς η ώρα, οπότε Άντωνη, να σας σταματήσω λίγο. Στην ημερήσια διάταξη ε, λεγόταν ότι ξεκινούσε η συνάντηση αυτή στις 4 και 20 και θα επαναληφθώ τώρα. Δεν ε, σας επιπλήττω, αλλά η ατζέντα είναι πάντα ευέλικτη. Αν κάτι συμβεί και κάτι συζητηθεί νωρίτερα, θα συζητηθεί νωρίτερα. Οπότε σας παρακαλώ και τους βοηθούς, σας παρακαλώ δεν μπορείτε να, να ενημερώνετε σίγουρα τα μέλη σας ότι τα πράγματα μπορεί να συζητηθούν λίγο νωρίτερα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό είμαι τόσο ευέλικτος, γι' αυτό δεν, δεν έχω κάνει και σχόλια μέχρι σήμερα. Γιατί ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκα είτε ξεκίνησε πιο νωρίς ή πιο αργά μια συνάντηση, πάντα περίμενα υπομονετικά τους άλλους. Νομίζω ότι ήταν μια καλή συνάντηση στο Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα. Ε, κάναμε διάφορες ε, συμβιβασμούς και εμείς από το ΕΛΚ ε, συμβάλαμε στο να έχουμε μια γνωμοδότηση έτσι και πρέπει να πω βέβαια το έργο της συναδέλφου κυρίας Κάλλας ήταν εξαιρετικό δεν δημιουργήθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα και νομίζω ότι αύριο θα στείλουμε ένα σαφές μήνυμα και αν εγκριθεί αυτή, αν εγκριθεί αυτή η έκθεση από αυτή την Επιτροπή και κατά την άποψή μου είναι σημαντικό να στείλει ΙΜΚΟ αυτό το μήνυμα ότι χρειαζόμαστε απόλυτη υλοποίηση των αγορών αυτών ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Το έχουμε συζητήσει μεταξύ συναδέλφων, μεταξύ πολλών ομάδων και όλοι έχουμε τους ίδιους στόχους. Επίσης πρέπει να δούμε τι γίνεται με τους φραγμούς που παρεμποδίζουν τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης. Οπότε εκεί θα βοηθήσουμε τις νέες τιμολογήσεις, θα επιτρέπουμε στους καταναλωτές να δημιουργούν οι ίδιοι ενέργεια και θα αναθέσουμε στην Κομισιόν να παρακολουθεί την υλοποίηση τη σύσταση 2012 για τους έξυπνους μετρητές και εμείς στο ΕΛΚ πιστεύουμε ότι είναι σημαντική για την υλοποίηση των ενεργειακών πολιτικών. Επίσης χρειαζόμαστε μεγαλύτερη σαφήνεια και διαφάνεια όσον αφορά το χειρισμό περίεργων ε, παραπώνων και τέλος πιστεύουμε ότι οι φόροι και τα τέλη που δεν σχετίζονται με την ενέργεια δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε λογαριασμούς ενέργειας. Ευχαριστώ λοιπόν που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία και ευχαριστούμε και πάλι για την έκθεση και πιστεύω ότι συμφωνούμε όλοι. Κάια, θα θέλατε να επανέλθετε. Δεν έχω να σχολιάσω πολλά. Όχι. Ίσως ένα πράγμα. Ε, λυπάμαι που ακούω ότι δεν μπορεί να υποστήριξει τη συμβαστική 2 το S&D γιατί εκεί προσπαθήσαμε εμείς να συμπεριλάβουμε και τις τροπολογίες τους. Ε, αλλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι Κατανοώ ότι η λέξη αγορά αποτελεί κόκκινη γραμμή για τους σοσιαλιστές, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να καταλάβουμε ότι για παράδειγμα στην αγορά των τηλεπικοινωνιών η απελευθέρωση οδήγησε σε μείωση των τιμών μεταξύ άλλων και, αύξησε και σε αύξηση των επενδύσεων στις αγορές αυτές. Οπότε ουσιαστικά σε όλες τις χώρες εκείνες όπου υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός έχουν πέσει οι τιμές. Οπότε αυτό ωφελεί και τους καταναλωτές. Οπότε δεν είναι ότι παραβλέπουμε το ζήτημα της ε, ενεργειακής ένδυας. Αλλά ταυτόχρονα είναι σαφές ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να επιτευχθεί ε, με την καταβολή επιπλέον φόρων και επιχορηγήσεων επιπλέον των τιμών τελικά κάποιος θα πρέπει να τα καταβάλει αυτά τα ποσά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Να κάνω μια πρόταση αν μου επιτρέπετε στη γραμματεία της Επιτροπής. Όταν αλλάζουμε την τα στοιχεία της ημερησίας διάταξης, επειδή κυκλοφόρησε μια νέα ημερησία διάταξη που κυκλοφόρησε την Πέμπτη ε, το μεσημέρι και την Τρίτη, και εκεί φαινόταν ότι μεταφερόταν η συζήτηση αυτή στις 4 και 20. Σας παρακαλώ όταν γίνονται τέτοιες αλλαγές να στέλνονται email στους εισηγητές και στους κοιόδης ώστε να διευκολύνουμε τα πράγματα γιατί ξέρω ο κόσμος ε, λαμβάνει πολλά email αυτό το email να έχει και τίτλο αλλαγή στην ημερήσια διάταξη σας ευχαριστώ παρόλα αυτά για την ευελιξία σας λοιπόν είναι δικό μου λάθος τώρα Υπήρξε ένα άλλο σημείο, μια ενημέρωση για τους τριμερείς διαλόγους, για τον τριμερή διάλογο, για την προσβασιμότητα, για στις ε, ιστοσελίδες ε, των δημοσίων οργανισμών και τη σχετική οδηγία και όπως φαίνεται ο εισηγητής είχε ζητήσει από μένα να διαβάσω την εκθέση αν συμφωνείτε λοιπόν να τη διαβάσω δεν έχω πρόβλημα να διαβάζω τις εκθέσεις εισηγητών αλλά παρακαλώ ειδοποιείτε τη γραμματεία εφόσον θέλετε να κάνω εγώ κάτι τέτοιο ώστε να το γνωρίζουμε μην ειδοποιείτε απλά το γραφείο μου, ειδοποιείτε και τη γραμματεία. Έκθεση λοιπόν για την οδηγία σχετικά με την προσβασιμότητα στις δημοσίων οργανισμών. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρώτη ανάγνωση, σε πρώτη ανάγνωση το κείμενό του 24 ε, Φεβρουαρίου. Ξεκίνησαν επίσημες διαπραγματεύσεις και στις 18 Δεκεμβρίου του 2015 ε, ξεκινήσαμε επίσημες ε, διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο στη διάρκεια της Ολλανδικής Προεδρίας. Υπάρχουν διάφορες ε, διαφορές μεταξύ των θέσεων των δύο θεσμικών οργάνων όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, τη φύση των διατάξεων ε, εφαρμογής ε, και κάποιες άλλες δράσεις όπως είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης. Είχαμε μια πρώτη διερευνητική συνάντηση στις 26 Ιανουαρίου, κάποιες τεχνικές συνεντήσεις και ο δεύτερος τριμερής διάλογος έγινε στις 2 Μαρτίου φέτος. Επί, παρότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές, Έχουμε σημειώσει προόδο και το Συμβούλιο έχει δείξει διάθεση να προσεγγίσει τη θέση του Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα όσον αφορά τα πρόσθετα μέτρα που θα εξασφαλίζουν ότι η οδηγία θα εφαρμόζεται επί τόπου και θα ε, επιτυγχάνει υψηλό βαθμό προσβασιμότητας των ιστοσελίδων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, επιβεβαίωσε το Συμβούλιο τη θετική του στάση απέναντι ε, στην πρόταση του Κοινοβουλίου για την χρήση σχολείων χρηστών σχετικά με την προσβασιμότητα και την διεύρυνση και την εφαρμογή προγραμμάτων αύξησης ευαισθητοποίησης. Το Συμβούλιο επίσης συμφωνεί με την ανάγκη να υπάρξει συνεπής προσέγγιση όσον αφορά την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι έχουμε πλησιάσει ο ένας τον άλλον ως προς τις θέσεις μας, είναι σαφές ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν δύσκολες και θα χρειαστεί ακόμη περισσότερο έργο για να καθοριστούν ε, οι τύποι των ιστοσελίδων και του περιεχομένου που θα συμπεριληφθεί και εκείνου που θα αποκλείεται από το πεδίο εφαρμογής του νομοθετήματος. Ο επόμενος τριμερής διάλογος αναμένεται να γίνει στις 26 Απριλίου του 2016 και επειδή γνωρίζω ότι λαμβάνουμε πολλά email για τις εφαρμογές θέλω να σας πω ότι σημειώνεται κάποια πρόοδος και σε αυτό το θέμα. Είχαμε κάποιες θετικές συζητήσεις στους τελευταίους τριμερείς διαλόγους για την ανάγκη κάλυψης και των εφαρμογών πέραν των ε, ιστοσελίδων. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα πέντε λεπτών, περιμένοντας την Κομισιόν, γιατί το τελευταίο θέμα μας είναι η παρουσίαση της Κομισιόν σχετικά με το θέμα των απαιτήσεων ε, προσβασιμότητας για προϊόντα και υπηρεσίες. Αλλά ο υπάλληλος της Κομισιόν, Μανουέλ Κελέν, δεν έχει έρθει ακόμη. Πέντε λεπτά διάλειμμα λοιπόν. Is this um, Director Manuela Gilling? Manuela Gilling βρίσκεται εδώ. Okay. Is this η κυρία Διευθύντρια Μανουέλα Γκέλινγκ βρίσκεται εδώ. Ε, ναι, λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε μαζί μας. Να σας υπενθυμίσω παρακαλώ και παρακαλώ να μεταφέρετε το μήνυμα στην Κομισιόν. Η ημερήσια διατάξη μας μερικές φορές ε, εξετάζει τα θέματα λίγο πιο γρήγορα, οπότε αρχίζουμε τη, κάποια συζήτηση νωρίτερα και πολλοί κόσμοι εδώ τώρα σας περίμενε για 15 λεπτά. Οπότε σας παρακαλώ καμιά φορά να έρχεστε και νωρίτερα γιατί μπορεί κάποια πράγματα να συζητηθούν νωρίτερα. Δεν μπορώ εγώ να προβλέψω πόσο χρόνο χρειάζομαι για το κάθε θέμα. Παρακαλώ, παρακαλέστε τους συναδέλφους σας να έρχονται λίγο νωρίτερα αν είναι δυνατόν διότι αλλιώς τα μέλη περιμένουν και η συνάντηση, η συνεδρίαση κάπως τελματώνει, δεν ρέει έτσι όμορφα όπως θα θέλαμε. Οπότε παρακαλώ να φτάνετε λίγο νωρίτερα. Λοιπόν, η πρόταση αυτή αφορά μια οδηγία για, την για τις απαιτήσει προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Η συγητής είναι ο ιδιαίτερα έμπειρος αντιπρόεδρος της Επιτροπής Γοσφόχ. Εδώ λοιπόν θα έχουμε μια παρουσίαση της πρότασης από την Κομισιόν. Μα ζήτησαν να εμπλακούν οι επιτροπέ αναφορών, μεταφορών και Απασχόλησης. Δεν έχουμε ε, συζητήσει ακόμα πότε όλα αυτά θα γίνουν ακριβώ, αλλά ανταλλάσσουμε μηνύματα τώρα με του Προέδρου των Επιτροπών αυτών. Οπότε τώρα δίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Εμμανουέλα Γκελάνγκ, να μα παρουσιάσει την πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Να ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση αυτή. Ξέρετε, εγώ είχα πριν από αυτή τη συνάντηση μια άλλη και μετά τρέξαμε για να έρθουμε στο κοινοβούλιο, αλλά όπω φαίνεται αργήσαμε. Σημειώνω τα όσα είπατε όμω, και θα τα μεταφέρω. Θα φροντίσουμε να ερχόμαστε νωρίτερα τι επόμενε φορέ. Ειδικότερα διότι αυτό εδώ το θέμα μας απασχολεί ιδιαίτερα και ε, θέλαμε, αναμένουμε με ανυπομονησία να παρουσιάσουμε αυτή την πράξη για την προσβασιμότητα. Έχουμε και εμεί διαφάνειες, τις οποίες μπορούμε να σας μοιράσουμε, αφού δεν μπορούμε να τις δείξουμε τώρα, εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον. Τι θα κάνουμε σήμερα. Θα απαντήσουμε μερικές ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, γιατί έχουμε προτείνει μια πράξη για την προσβασιμότητα, ποιος επωφελείται από αυτήν, τι καλύπτει η πράξη αυτή, τι δεν καλύπτει η πράξη αυτή, τα ζητήματα της αναλογικότητας και της επικουρικότητας και το χρονοδιάγραμμα που αφορά την πράξη αυτή. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, οι λόγοι για τους οποίους εξετάζουμε μια τέτοια πράξη προσβασιμότητας είναι μεταξύ άλλων οικονομική. Πρώτα απ' όλα πρέπει να βελτιώσουμε τη σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς για προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτό θέλουμε να το επιτύχουμε εναρμονίζοντας ε, τους διαφορετικούς κανόνες προσβασιμότητας και διασφαλίζοντας την ελεύθερη κυκλοφορία των προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, διευκολύνοντας έτσι το έργο της βιομηχανίας ε, και ε, βοηθώντας να οδηγηθούμε σε υγιή ανταγωνισμό, πιο προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες σε πιο ανταγωνιστικές τιμές. Η Υπάρχει μια αγορά. Αυτή η πράξη για την προσβασιμότητα θα επηρεάσει θετικά 18 εκατομμύρια ε, ανάπηρους ανθρώπους, περίπου το 20% επίσης του ευρωπαϊκού πληθυσμού που γυράσκει και που έχει περιορισμούς ε, κινητικούς κοινωνία μας ψηφιοποιείται όλο και περισσότερο. Σε ολόκληρο τον κόσμο λαμβάνονται μέτρα βελτίωση της προσβασιμότητας των τεχνολογιών πληροφοριών ε, ε, και επικοινωνιών, οπότε πρέπει να γίνουμε ανταγωνιστικοί στο παγκόσμιο στερέωμα. Ποιε είναι τώρα οι νομικές υποχρεώσεις, Ποια, συγγνώμη, ποιες είναι οι νομικές αιτίε, Πρώτα απ' όλα έχουμε νομικές υποχρεώσεις. Η Συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των ανθρώπων με Αναπηρίες ε, τέθηκε σε ισχύ το 2011 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ένωση ίδια και οι 25 κράτη-μέλη έχουν επικυρώσει τη σύμβαση και τρία βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης της διαδικασίας επικύρωσης. Η συνθήκη ε, θέτει υποχρεώσει ε, για τα μέλη για εξασφάλιση της προσβασιμότητας στον τομέα των μεταφορών και των, της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Έτσι λοιπόν πρέπει να βελτιώσουν τη σχετική νομοθεσία τα κράτη-μέλη. Αν δεν υπάρχει συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα οδηγηθούμε σε διαφορές και κατακρεματισμό των νομοθεσιών στην εσωτερική αγορά. Η πράξη για την προσβασιμότητα φυσικά δεν αποτελεί τη μόνη απάντηση για την άρση του κατακρεματισμού, ωστόσο περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαιτεί η συνθήκη τα οποία εφόσον υιοθετηθούν και εφαρμοστούν θα βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να σημειώσουν πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση του άρθρου 9 της σύμβασης που περιλαμβάνει την υποχρέωση προσβασιμότητας. Ποιο επωφελείται από την άρση των εμποδίων. Πρώτα απ' όλα η βιομηχανία είναι σαφές, η παραγωγή, η παροχή υπηρεσιών, οι κοινέ ε, απαιτήσει προσβασιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα διευκόλυναν και θα απλούστευαν το έργο τους και θα τους παρέχαν ασφαλεία δίκαιότητα τα προϊόντα τους πληρούν ε, τις ε, προϋποθέσεις προσβασιμότητα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι θα επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία φυσικά και η καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς θα ήταν μια απόρρια των πλέον προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών και αυτό θα ωφελήσει και τους ανθρώπους με αναπηρίες ή τους ε, γυρότερους ε, πολίτες ε, προσφέροντας τους περισσότερες επιλογές, καλύτερη ποιότητα και καλύτερες τιμές. Επιπροσθέτως ε, όλοι οι υπόλοιποι θα υποφεληθούν από όλο αυτό. Είμαι βέβαιο ότι θα προσπαθήσετε ε, θα έχετε προσπαθήσει να διαβάσετε μια οθόνη έχοντας ξεχάσει τα γυαλιά σας ή καμιά φορά δεν θα μπορούσατε να δείτε την οθόνη πάνω σε ένα ATM όταν πέφτει ο ήλιος πάνω ή όταν προσπαθείτε να ακούσετε μια ανακοίνωση σε έναν πολύβο σιδηροδρομικό σταθμό. Αλλά πιστεύω ότι και αυτοί που θα υποφεληθούν ιδιαίτερα θα είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές ουσιαστικά είναι οι πλέον ευάλωτες στον κατακαιρματισμό της νομοθεσίας. Έχουν περιορισμένους πόρους, δεν μπορούν εύκολα να μάθουν και να εφαρμόσουν τους πιθανότατα 27-28 διαφορετικούς κανόνες του κάθε κράτους μέλους και η συμμόρφωση λοιπόν με ένα μόνο σύνολο κανόνων είναι κάτι αναπόφευκτο. είναι ε, τεράστιο πλεονέκτημα, έκτημα αντί να χρειάζεται κανείς να συμμορφώνεται με διαφορετικά, ε, διαφορετικούς κανόνες ε, διαφορετικών κρατών μελών. Ειδικότερα λοιπόν για τις μικρές εταιρείες η δυνατότητα αυτή η πρόσβαση σε όλες τις αγορές αποτελεί σίγουρα ένα πλεονέκτημα. Τι καλύπτει η, πράξη, η ευρωπαϊκή πράξη προσβασιμότητας. Να αναφέρω πρώτα απ' όλα καθαρά ότι αυτή είναι μια πρωτοβουλία φιλική προς τους χρήστες που χρησιμοποιεί όπως γνωρίζετε τα καθιερωμένα εργαλεία της εσωτερικής αγοράς βασίζεται σε υπάρχουσες πρακτικές και δομές. Κατά βάση έχει δύο σκέλη. Το ένα θέτει υποχρεώσεις προσβασιμότητας για συγκεκριμένο αριθμό προϊόντων και υπηρεσιών που υφίστανται ρυθμίσεις και είναι πιθανό να ε, ε, υποστούν και περισσότερες ρυθμίσεις ενώ έχουν εντοπιστεί ως προϊόντα και υπηρεσίες κλειδί για πολίτες με αναπηρίες. Το δεύτερο σκέλος της πράξης χρησιμοποιεί ακριβώς τις ίδιες απαιτήσει για τη διευκρίνηση του νοήματος της προσβασιμότητας στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που ήδη περιλαμβάνει σχετικές διατάξεις. Αναφέρομαι εδώ παραδείγματι στην ε, οδηγία περί δημοσίων συμβάσεων που πρέπει να είναι προσβάσιμη ο κανονισμός για τα διορθωτικά ταμεία που απαιτεί να λαμβάνεται υπόψη προσβασιμότητα κατά την υλοποίηση των ταμείων και την προετοιμασία τους. Αλλά καμία από αυτές τις δύο πράξεις δεν περιγράφει επακριβώς την προσβασιμότητα. Η απαιτήσει λοιπόν προσβασιμότητας αυτής της οδηγίας θα χρησιμοποιηθούν για αυτόν ακριβώς τον αρισμό σε αυτές τις περιπτώσεις. Τι προτείνεται μέσω της πράξης αυτής. Καταρχάς η πράξη αποτελεί ένα πλαίσιο για την προσβασιμότητα στην Ευρώπη. Χρησιμοποιεί απλές διαδικασίες αφήνοντας περιθώριο για καινοτομία και μελλοντικό έλεγχο καθιστά υποχρεωτικές ορισμένες λειτουργικές απαιτήσει για τα επιλεγμένα προϊόντα και τις υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα παρέχει την δυνατότητα θελοντικά εναρμονισμένων προτύπων, ώστε να καλύπτεται ε, η απαιτήση συμμόρφωσης ε, και να διευκολύνεται η υλοποίηση των απαιτήσεων. Οι ίδιοι οικονομικοί φορείς όμως θα είναι εκείνοι που θα αξιολογούν ε, και θα αποφασίζουν κατά πόσο ένα προϊόν ή μία υπηρεσία συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές και αφήνει να χρησιμοποιούν τη μηχανισμοί των αγορών για να ελέγχεται τακτικά η συμμόρφωση και παρέχει και μηχανισμούς επιβολής του νόμου για τους καταναλωτές οι οποίοι μπορούν να απαιτήσουν με αυτόν τον τρόπο τη συμμόρφωση. Έτσι διασφαλίζει ότι αφού ε, συμμορφούνται με τι προδιαγραφέ τα προϊόντα και μπορούν να κυκλοφορήσουν ελεύθερα σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά. Όλα αυτά βάσει καλά καθιερωμένων διαδικασιών και μηχανισμών γνωστών στην εσωτερική αγορά. Τώρα κάτι πιο σημαντικό ακόμα. Τι δεν κάνει η πράξη αυτή. Πρώτα απ' όλα δεν περιγράφει σε επίπεδο τεχνικών λεπτομεριών πώς ε, καθίσταται συμβατό ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Για παράδειγμα, όσον αφορά τον, την ποσότητα, λέει ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος έλεγχος ε, ε συγγνώμη, έντασης ήχου, για παράδειγμα. Ε, δεν λέει όμως αν πρέπει να υπάρχει κουμπί περιστρεφόμενο ή άλλο για τη ρύθμιση του ήχου. Δεν ορίζει υποχρεώσεις για όλους τους ε, κατασκευαστές και παρόχους υπηρεσιών ε, θέτει, προβλέπει κάποιες υποχρεώσεις μόνο για αυτούς που έχουν επιλεγεί βάσει μιας ε, διαδικασίας επιλογής που πραγματοποιήθηκε κατά την εκτίμηση δικτύπου. Δεν επιβάλλει μη ρεαλιστικές ή επαχθείς υποχρεώσεις. Υπάρχουν διασφαλίσεις όλες τις διατάξεις αυτές δεν τροποποιεί τομεακή νομοθεσία που υπάρχει ήδη περί προσβασιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά μάλλον συμπληρώνει και ισχύει τους υπάρχοντες κανόνες. Να σας πω τώρα δύο λόγια για την εκτίμηση δικτύπου. Η εκτίμηση δικτύπου έχει συνταχθεί πολύ σωστά και έχει ολοκληρωθεί εντός του 2013 καλύπτει 80% του των υπηρεσιών και το 70% του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Επίσης, περιλαμβάνει στοιχεία από έρευνες που έχουν γίνει από δίκτυο πανεπιστημιακών εμπειρογνωμόνων, που καλύπτει κάθε κράτος μέλος, δίνοντας έτσι μια εικόνα για την νομοθετική κατάσταση για βασικά προϊόντα και υπηρεσίες. Επίσης, είχαμε συμμετοχή και συμβολή από διάφορες διαβουλεύσεις που βοήθησαν στο να εντοπίσουμε προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και ε, τα εργαλεία της εσωτερικής αγοράς που θα είναι τα πιο χρήσιμα. Η αξιολόγηση αντικτύπου αναλύει διάφορες επιλογές, ε, πιο ελαφρές, νομοθετικές, και εν τέλει απορρίπτει πέντε επιλογές γιατί θεωρήθηκαν μη ρεαλιστικές. Ενώ στηρίζει τέσσερις άλλες επιλογές που αναλύονται με λεπτομέρειες. Πώς τώρα αυτή η πρόταση συνδέεται με την παλιότερη ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία. Καταρχά, όπως ανέφερα και προηγουμένως, για να ανταποκριθ για να αντιστοιχιστεί η ζήτηση με την ε, προσφορά ζητάμε τα ίδια εργαλεία ε, για τους ρυθμιστές και τους ε, κρατικούς προμηθευτές όταν αγοράζουν, πουλούν προϊόντα και υπηρεσία. Οι οικονομικοί φορείς που θα καταστήσουν εύκολα στη διάθεση, σε διάθεση εμπορική τα προϊόντα θα πρέπει να είναι προσβάσιμοι και για τις δημόσιες υπηρεσίες. Υπάρχει ο όρος της προβασιμότητας, αλλά δεν ορίζεται. Οπότε στην πράξη θα δείτε ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που εξετάζεται είναι η οδηγία για τις εκατοικές προμήθειες, οι κανονισμοί που διέπουν τα διαρθρωτικά και τα επενδυτικά ταμεία, ε, οι δημόσιες υπηρεσίες ε, ε, επιβατικών μεταφορών και εδώ δεν τροποποιείται καμία νομοθεσία ούτε κάποιο πεδίο εφαρμογής, αντίθετα στηρίζει και διευκολύνει την εφαρμογή των υφιστάμενων οδηγιών μέσω των απαιτήσεων προσβασιμότητας. Σύντομα θα ήθελα να σας παρουσιάσω πώς αυτή η πράξη συνδέεται με δύο, άλλες, ε, ε, με δύο άλλα νομοθετήματα. Το ένα είναι η οδηγία του άρθρου 19. Τα δύο αυτά μέσα είναι παραπληρωματικά, αλλά επιδιώκουν διαφορετικούς στόχους και έχουν και διαφορετικές νομικές βάσεις. Το άρθρο, η οδηγία του άρθρου 19 καταπολεμά τις διακρίσεις και εστιάζει στους ανθρώπους. Αυτή η πράξη, για ποια οδηγία είπατε, την οδηγία άρθρου 19. Είναι η οδηγία ε, κατά των διακρίσεων. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. So, um, as I was saying, the anti-discrimination Όπως έλεγα λοιπόν, η οδηγία κατά των διακρίσεων καταπολεμά τις διακρίσεις και εστιάζει στους ανθρώπους, ενώ η πράξη για την προσβασιμότητα στόχο έχει να βελτιώσει την πρόσβαση στην νέα αγορά χρησιμοποιώντας την εναρμόνιση. Αρχίζει λοιπόν εξετάζοντας προϊόντα και υπηρεσίες. Βεβαίως και οι δύο συμβάλλουν στην εφαρμογή της σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ανθρώπων με ε, δυσκολίες ή με ειδικές ανάγκες, αλλά έχουν διαφορετικούς στόχους. Κάτι ακόμα θα πρέπει να έχουμε υπόψη και αφορά την οδηγία για την πρόσβαση στο δίκτυο. Ακόμα ένα μέσο που είναι υποδιαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή. εστιάζουμε στην πρόσβαση στα, στους διάφορους ιστότοπους. Όταν ε, σχεδιάστηκαν αυτές οι οδηγίες δεν υπήρχε επικάλυψη και η πλήρη συμβατότητα ανάμεσα στα μέσα έχει εξασφαλιστεί, οπότε ε, καθώς προχωράει η συζήτηση ε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πως η συνοχή και ο συντονισμός ανάμεσα στις δύο πράξεις αυτές θα διατηρηθούν. Να πω ε, δύο λόγια για την αναλογικότητα και την επικουρικότητα. Καταρχάς αυτή η οδηγία εστιάζει στην αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουμε αντιμετωπίσει. Είναι ευέλικτη και στοχοθετημένη. Και να σας εξηγήσω γιατί. Είναι ε, ε, στοχοθετημένη γιατί μιλά μόνο για εκείνα τα προϊόντα και τις παραγωγές όπου υπάρχουν αποκλίνουσες νομοθεσίες και εκεί όπου υπάρχει μια ευρωπαϊκή διάσταση. Γι' αυτό τον λόγο, όταν εξετάσει κανείς την πράξη, θα δείτε ότι το περιβάλλον γύρω από το οποίο κινούνται και παρέχεται η υπηρεσία ε, αναφέρεται μέσω μιας ρήτρα διευκόλυνσης. Δηλαδή το κρατός μέλος θα έχει την επιλογή αν θα χρησιμοποιήσει τις ίδιες απαιτήσεις προσβασιμότητας ή όχι. Τα, οι απαιτήσει προσβασιμότητας ισχύουν μόνο για νέα προϊόντα αλλά και για την παροχή νέων υπηρεσιών Οπότε δεν υπάρχει απέταση για αναδρομική ισχύ για προϊόντα και υπηρεσίες. Η απέτηση προσβασιμότητας ορίζεται σε λειτουργικό επίπεδο. σα το έδωσα το παράδειγμα της έντασης του ήχου. Επίσης έχουμε εισάγει ε, μια ελαφριά ε, αξιολόγηση συμμόρφωσης, δηλαδή μια δήλωση μια υπεύθυνη δήλωση και αυτό για να διευκολύνουμε τους οικονομικούς φορείς και για να εξασφαλίσουμε την αναλογικότητα των υποχρεώσεων. Υπάρχουν δύο ρήτρες ασφαλείας που ήδη ανέφερα. Η μια περιορίζει τους υποχρεώσεις στο βαθμό που δεν επιβάλλουν δυσανάλογο φόρτο και η δεύτερη δεν απαιτεί αλλαγή στη θεμελιώδη φύση του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Για παράδειγμα, η υποχρέωση της e-books απαιτείται να περιλάμβουν ε, χαρακτηριστικά προσβασιμότητα στους ηλεκτρονικούς φακέλους, ας πούμε, όσον αφορά τη δομή και την πλοήγηση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αλλάξει το προϊόν, ώστε να είναι ένα βοηθητικό βιβλίο με braille ή με κωδικοποιημένες φωνές. Πράγμα που αλλάζει τελείως τη φύση του ηλεκτρονικού βιβλίου. Βεβαίω οι οικονομικοί φορεί θα πρέπει να αιτιολογήσουν και να εξηγήσουν την αξιολόγησή του, κοινοποιώντα τι αρμόδιε αρχέ και θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι από αυτέ τι αρμόδιε αρχέ. Οπότε υπάρχει μια προσεκτική ισορροπία ανάμεσα στην ευθύνη και την εμπιστοσύνη που έχει τοποθετηθεί στους οικονομικούς ε, ε, φορείς και τους ελέγχους που πρέπει πρέπει να προβαίνουν οι αρμόδιες αρχές κάθε φορά χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή. Έχουμε δει δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύω ε, της ε, περίοδου μεταγραφής Έχουμε δει ότι η αρχή της ισχύω ε, θα είναι έξι χρόνια μετά από την έγκριση και η Κομισιόν θα πρέπει να υποβάλει την πρώτη της έκθεση σε σχέση με την εφαρμογή της οδηγίας πέντε έτη μετά από την ημερομηνία εφαρμογής της. Η έκθεση αυτή έχει στόχο να εξασφαλίσει ότι στη διάρκεια της εφαρμογής της η οδηγία θα εξακολουθήσει να εξυπηρετεί τους στόχους της. Αν κατακλείδη θα ήθελα να σας δώσω μια γενική εικόνα των απόψεων των εμπλεκομένων φορεών όπως τις έχουμε συλλέξει Συχνά βεβαίως ακούσαμε εσάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ζητάτε από την Κομισιόν να δράσει και να υιοθετήσει την πράξη περί την, το νομοθέτημα μάλλον για την ε, προσβασιμότητα, γιατί αυτό θα επηρεάσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Επίσης, έχουμε ακούσει την ε, απόψεις της ε, ομάδας υψηλού επίπεδου για τη σκοπιμότητα, για το δυναμικό που έχει η πρόταση αυτή να βελτιώσει συγκεκριμένα τις δυνατότητες πρόσβασης. Από τον ε, κλάδο ακούσαμε ότι ανησυχεί σε σχέση με τον κατακαιρματισμό και την απόκληση μιας νομοθεσίας που στόχο έχει Ε, όπου στόχο έχει να εφαρμοστούν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Ωστόσο, θα πρέπει, ε, αποδέχονται ότι είναι πολύ στοχοθετημένοι, ότι αφορά πολύ συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Τα προϊόντα ε, έχουν να κάνουν με τους υπολογιστές, τη τηλεφωνία, τα μηχανήματα ATM, τα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων, ελέγχου εισιτηρίων, υπηρεσίες τηλεφωνίας, μεταφορών, site οπτικοακουστικών μέσων, μάλλον οπτικοακουστικά μέσα και πέρα από αυτά, από αυτούς τους καταλόγους προϊόντων και υπηρεσιών θα παραμένουν πάντοτε προϊόντα και υπηρεσίες που τα άτομα με δυσκολίες θα τα χρειάζονται και για τα οποία τα οποία δεν εμπίπτουν εδώ, αυτά παραμένουν στην ευθύνη των κατών μελών. Ωστόσο, θα πρέπει να πω ότι οι άνθρωποι με ειδικέ ανάγκε έχουν πολλέ προσδοκίε από, από ε, αυτό το νομοθέτημα δεδομένων των ε, δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει για να εξασφαλίσουμε την προσβασιμότητα υπό την σύμβαση. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτή η σύμβαση είναι ένας τρόπος συνεργασίας ώστε να εφαρμοστεί κάνοντας την καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων, των λιγοστών πόρων που υπάρχουν στην Ευρώπη και έτσι να βελτιώσουμε την ενιαία αγορά και για αυτούς τους ανθρώπους. Ευχαριστώ. Ο Ρόμπερτ. Ευχαριστώ Βίκη, ευχαριστούμε κύριε Διευθύντρια για αυτή την πολύ ολοκληρωμένη περιεκτική παρουσίαση αυτού του πολύ όμορφου κειμένου, πολύ όμορφου ε, νομοσχεδίου. Πιστεύω ότι η πρότασή σας είναι σαφής, έχει συνοχή. Αλλά επειδή πρόκειται για ένα ευαίσθητο θέμα, ε, είναι και πολύπλοκη η πρόταση αυτή. Οπότε χρειάζεται να μελετήσουμε διεξοδικά το κείμενο αυτό τις επόμενες εβδομάδες. Το θέμα δεν είναι απλά να βελτιώσουμε τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, όπως πολύ συχνά λέμε εδώ. Το θέμα είναι να αυξήσουμε την εσωτερική αγορά να πράξουμε έτσι ώστε να μπορέσει να ενταχθεί ολοκληρωμένα ε, σε έναν τομέα όπου σήμερα υπάρχουν περιορισμοί, και καινοτομίες που καθυστερούν και έτσι λοιπόν σε τελική τι προσπαθούμε να πούμε όλοι μας και εσείς και εμείς. Το πρώτο είναι ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες δεν πάβουν να είναι καταναλωτές. Καταναλωτές με τα ίδια δικαιώματα. Νομικά αλλά όχι τα ίδια δικαιώματα όσον αφορά την πρόσβαση στα προϊόντα. Διότι ορισμένα προϊόντα δεν τους είναι προσβάσιμα πολύ απλά, διότι τα προϊόντα αυτά δεν ε, έχουν συναντήσει επαρκή αγορά για να αναπτυχθούν, κυρίως λόγω του κατακρεματισμού των νομοθεσιών μεταξύ των κρατών μελών. Παρομοίως, οι επιχείρησεις που κατασκευάζουν τα προϊόντα αυτά ή τα παράγουν, αν ε, έχουν ένα ενιαίο πλαίσιο θα έχουν μια ευρύτερη αγορά και θα μπορούν να δραστηριοποιούνται ακόμη περισσότερα για να ε, εξυπηρετήσουν τα οικονομικά του συμφέροντα. Όταν λέμε 120 εκατομμύρια είναι οι Ευρωπαίοι που θα μπορούσε να αφορά αυτό το σχέδιο οδηγία, δηλαδή ουσιαστικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχεδόν ένα στου τέσσερι. Ένα στου τέσσερι. Δεν μιλάμε δηλαδή για μια μικρή ξεχασμένη ομάδα. Μιλάμε για ένα σημαντικό κομμάτι της εσωτερικής αγοράς. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με κάτι ε, και κάνατε πολύ σωστά που διαλέξετε την οπτική γωνία της εσωτερικής αγοράς. Διότι αυτή η εσωτερική αγορά ε, καλύπτει τις οικονομικές ανάγκες ε, και μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη εδώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ίσως και να την φέρει πιο μπροστά από άλλες περιοχές του κόσμου για τέτοια θέματα που θα είναι θέματα που θα μας απασχολήσουν στο μέλλον. Η Βίκη μας υπενθύμισε προηγουμένως ότι πολλές επιτροπές ε, ενδιαφέρονται για το θέμα και χαιρόμαστε γι' αυτό ε, και είμαστε βέβαιοι ότι θα καταφέρουμε να βρούμε έναν τρόπο συνεργασίας επικοδομητικά μαζί με συναδέλφους άλλων επιτροπών. Λοιπόν, όπως είπατε, οι προσδοκίες είναι μεγάλες και η στιγμή είναι πρόσφορη. Εδώ και καιρό περιμέναμε να ακούσουμε κάτι φιλόδοξο. Δεν ξέρω αν άξιζε τον κόπο να περιμένουμε τόσο καιρό, αλλά σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα είναι εδώ πλέον και είναι σημαντικό, όπως διαπιστώνουμε. Επίσης πιστεύω δικαίως επικεντρώνεστε στο ψηφιακό τομέα το κείμενο αυτό, ξέρετε, θα μπορούσε να ενταχθεί αυτούσιο σε μια δέσμη μέτρων για την ψηφιακή αγορά ε, λόγω των προϊόντων που επιλέξατε που ανήκουν σε μεγάλο βαθμό στην ψηφιακή αγορά. Από την άλλη, εξετάζοντας ε, τις διάφορες δυναμικές εντός των καταναλωτών στην Ευρώπη, σε ε, όλον το μυαλό έρχεται η δημογραφική γύρανση. Δηλαδή άνθρωποι που χωρίς αναπηρία συνεχίζουν να είναι καταναλωτές αλλά με μειωμένες δυνατότητες λόγω ηλικίας ή λόγω χρόνων ασθενειών. Δηλαδή άνθρωποι πλέον χωρίς αναπηρίες ε, παρόλα αυτά επιζούν για πάρα πολλά χρόνια, ζουν πάρα πολλά χρόνια ε, αλλά λόγω κάποιες ασθένειας ε, έχουν κάποιο περιορισμό κινητικότητας αλλά δεν πάβουν να είναι καταναλωτές για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Ε, καλά κάνετε και υπενθυμίστε τη συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών που υποχρεώνει τα κράτη να δράσουν. Διαφορετικά υπήρχε κίνδυνος ε, να κινηθούμε προς την αντίστροφη κατεύθυνση της, ε, από αυτή της ενίας αγοράς. Κάτι ανεπιθύμητο. Οπότε χρειάζεται απόλυτη σαφήνεια για να μην αρχίσουμε να όπως το χωρούμε, να, να όπως το δρομούμε. Να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις αρχικές, έτσι για να ξεκινήσουμε μαζί τη συνεργασία μας. Κάποιες από αυτές τις ερωτήσεις ε, τις έχετε ήδη απαντήσει, ε, απλά να τις ξαναθέσω εγώ. Λοιπόν, είπατε πολύ σωστά ότι αυτή η πρόταση νομοθετικής πράξης αφορά μόνο ορισμένους τομείς προτεραιότητας που έχετε επιλέξει και όπως σας είπα και εγώ παρατήρησα ότι χαρακτηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από τα ψηφιακά, ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες ε, κάτι πολύ επίκαιρο αλλά η ερώτησή μου είναι πώς τα επιλέξατε πώς επικεντρωθήκατε σε συγκεκριμένους τομείς για ποιο λόγο περιοριστήκατε σε αυτά γιατί δεν επεκταθήκατε λίγο παραπέρα γιατί δεν είδατε τέτοια ανάγκη να επεκταθείτε λίγο παραπέρα από τον κατάλογο αυτών των προϊόντων που αναφέρετε στην πρόταση διότι σε τελική ανάλυση γιατί όχι αφού ασχοληθήκατε, που ασχοληθήκατε με την εσωτερική αγορά ε, και η οποία αφορά και τους καταναλωτές με περιορισμούς ε, κινητικότητας ε, θα έλεγε κανείς δεν είναι μόνο οι τραπεζικές υπηρεσίες ούτε μόνο οι ψηφιακές υπηρεσίες και κάποια προϊόντα υπάρχουν ένα σώρο άλλα πράγματα οπότε θα ήθελα να καταλάβω τη λογική σας τη λογική με την οποία περιοριστήκατε σε αυτό το πεδίο δεύτερον το κείμενο είναι φιλόδοξο όσον αφορά την προτινόμενη μέθοδο εδώ δεν βρισκόμαστε σε περίπτωση αυτορύθμισης, ε, δεν λέμε ότι όλα θα αυτορυθμιστούν από μόνα τους, ούτε βρισκόμαστε σε φάση αυταρχικής ε, τυποποίησης. Είμαστε σε κάτι που συντονίζεται με το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Αποτελεί συνέχεια του κειμένου για την ασφάλεια των προϊόντων ε, που είχε η την Βίκη και στο οποίο εργαστήκαμε πριν λίγο καιρό στην Επιτροπή μας. Ε, ξέρετε και όπως βλέπουμε είναι πολύ έξυπνο το να δουλεύει κανείς έτσι. Είναι μια από τις πτυχές της βελτίωσης της νομοθεσίας. Ε, ταυτόχρονα όμως ε, αντιλαμβανόμαστε ότι κάνει να φαίνεται κάτι άλλο πολύ σημαντικό ότι οι αρχές επιτήρησης των αγορών που είναι οι θεματοφύλακες ελέγχουν κατά πόσο βρήκαμε σωστό συμβιβασμό, σωστό κοινό τόπο, αυτές θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Πιστεύετε λοιπόν ότι αυτέ οι αρχές επιτρήσει τη αγορά σήμερα είναι σε θέση να διδραματίσουν τέτοιο ρόλο. Διότι το όλο εγχείρημα θα είναι πολύ πιο περίπλοκο από ό,τι φανταζόμαστε. Ποια είναι η απαντήσή σας γι' αυτό τώρα για τι προθεσμίε. Το αναφέρατε ε, επιτρέψτε μου έτσι να εμβαθύνω λίγα στις ερωτήσεις μου. Ξέρετε, η προστίκη των χρονοδιαγραμμάτων και προθεσμιών ε, θα δημιουργήσει καθυστερήσεις. Ε, λέτε δύο χρόνια μέχρι να μεταφερθεί η οδηγία, έξι χρόνια για να υιοθετήσουν τα κράτη-μέλη τα μέτρα εφαρμογής και μεταφοράς και μετά ο απολογισμός πέντε χρόνια μετά. Ξέρετε, έτσι φτάνουμε στο 2028 με ένα γρήγορο υπολογισμό για την τελική υλοποίηση εφόσον νομοθετική πράξη υιοθετηθεί το 2014. Ξέρετε, όταν 2028 είναι μια μακρινή ημερομηνία. Πόσο που τα προϊόντα στα οποία εσείς δίνετε εδώ προτεραιότητα είναι προϊόντα τα οποία κινούνται πάρα πολύ γρήγορα. Ε, θυμηθείτε την, επανάσταση, την ψηφιακή επανάσταση και πώς άλλαξε τα πράγματα το να έχουμε λοιπόν μια τέτοια καθυστέρηση δεν αποτελεί κάποια αντίφαση. Για παράδειγμα, για προϊόντα όπως τα smartphone, τα έξυπνα τηλέφωνα, δεν θα έπρεπε να προβλέψουμε μικρότερες προθεσμίες. Δεν πέφτουμε σε κάποιο είδος ασάφεια όσον αφορά αυτές τις καθυστερήσεις. Τώρα, ε, για τις υπηρεσίες είναι σαφές ότι τα λογισμικά και τα hardware πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στην όλη κατάσταση αλλά επίσης κάτι άλλο πρέπει όταν ε, υπάρχει πρόσβαση σε τέτοια λογισμικά ή μηχανήματα εντός ενός κτηρίου πρέπει και το κτίριο να είναι προσβάσιμο. Εσείς λοιπόν εδώ έχετε υιοθετήσει μία προσέγγιση όχι υποχρεωτική αλλά ε, προαιρετική. Τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό, υπάρχει περίπτωση να καταλήξουμε σε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Όταν τα κράτη-μέλη ε, δεν χρειάζεται υποχρεωτικά να εφαρμόσουν ε, όλες αυτές τις διατάξεις και στο περιβάλλον και στα κτίρια. Τέλος, ε, εγκρίνω απόλυτα το ότι αναφέρεται λειτουργικές απαιτήσει για τα προϊόντα αλλά σε καμία περίπτωση δεν λέτε πώς θα υλοποιηθούν αυτές οι απαιτήσει από τους βιομήχανους, από τους οικονομικούς φορείς. Εδώ με βρίσκεται απόλυτα σύμφωνο. Αυτό θα δώσει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να καινοτομήσουν, να δημιουργήσουν, να δώσουν απαντήσεις ε, βάσει των δικών τους ε, μέσων, μηχανικών, ε, σχεδιαστών. Αυτό θεωρώ είναι εξαιρετικά σημαντικό. Επίσης τίθεται το πολύ ενδιαφέρον ερώτημα του καθεστώτος εξαίρεσης, ελάφρυνσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 Όλα αυτά είναι επίσης ιδιαίτερα ευθύ και πιστεύω πολύ σημαντικά. Οπότε το ερώτημά μου είναι το εξή. Πώς θα καταφέρουμε να επιτύχουμε μια σωστή ισορροπία εκεί. Τι θα κάνουμε ώστε Δηλαδή που θα βάλουμε το όριο. Εάν συμπεριλάβουμε ένα περιθώριο ελιγμών όπως πρέπει, μήπως αυτό είναι τον κίνδυνο του να προσθέσουμε υπερβολικά μεγάλο περιθώριο με αποτέλεσμα τελικά ανεπαρκή προσβασιμότητα. Θα δω σε αυτές τις ερωτήσεις. αντιλαμβάνομαι ότι οι απαντήσει δεν είναι εύκολες. Ίσως να είναι και κάτι το οποίο θα χρειαστεί να σκεφτείτε πρώτα. Ε, αυτή να υπάρχει κάποια ρήτρα αναθεώρησης ίσως για να δούμε πώς θα αναθεωρηθεί αυτή η οδηγία. Τώρα και επανερχόμενος σε αυτά που είπε η δίκη προηγουμένως, όλα αυτά πρέπει να τα δούμε σαν ένα ανοικό κλείσμα των ματιών. Ξέρετε, όταν κάποιος υποφέρει από κάποια κινητικότητα ή κάποια αναπηρία, οι προθεσμίες και τα χρονοδιαγράμματα είναι πολύ δύσκολα πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε αυτό το κείμενο για την προσβασιμότητα και τελικά μας θυμίζετε ότι η προσβασιμότητα, μιλώντας γι' αυτό, μας λέτε ότι προσβασιμότητα σημαίνει να βάλουμε και τους αυτούς μας στη θέση αυτών των ανθρώπων. Και όταν διάβασα εγώ τον κατάλογο των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο δικό σας ε, κείμενο, μιλάτε για πολλά ψηφιακή, ψηφιακά προϊόντα, ε, για το πώς ε, ε, αντισταθμίζει κανείς τις ελλείψεις μιας αίσθησης μέσω μιας άλλης αίσθησης. Δεν θα έπρεπε λοιπόν στον ορισμό προσδοσμού να μιλάμε και περί ταχύτητας. Άνθρωποι με κάποιους τέτοιους περιορισμούς δεν μπορούν να παρακολουθήσουν, να ακολουθήσουν τις ταχύτητες αυτών των νέων τεχνολογιών. Οπότε η προσβασιμότητα θα πρέπει να παρέχει και τη δυνατότητα ε, να υπάρχουν ταχύτητες σε τέτοια προϊόντα χαμηλότερες από αυτές που υπάρχουν για ανθρώπους χωρίς λειτουργικά προβλήματα και που τρέχουν συνέχεια. Τρέχουν συνέχεια μερικές φορές τόσο πολύ που πολλές φορές δεν καταφέρουν αυτό στην ώρα τους. Ναι, συγγνώμη που ο, ο κύριος Χάνιμαν, ε, κυρία Λί, σήμερα διότι βρίσκεται στην ε, συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτισμού που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να μεταφέρω εκ μέρους της τα εξής. Σας ευχαριστούμε για αυτό το νομοθετικό κείμενο. Είναι ένα σημαντικό κείμενο για 18 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση μεγαλύτερη προσβασιμότητα θα δώσει μεγαλύτερες δυνατότητες σε εκατομμύρια ανθρώπους. Επιπλέον, με περισσότερες ψηφιακές δυνατότητες η προσβασιμότητα μπορεί να γίνει πιο διαθέσιμη και πιο ε, οικονομικά προσιτή σε μια σειρά από τομείς. Θα συμβάλλει στην λειτουργία της ενιαίας αγοράς μέσω εναρμονισμένων κριτηρίων για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά θα δημιουργήσει και κόστος για τις επιχειρήσεις και εκεί θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το κόστος αυτός δεν θα είναι υπερβολικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης θα ήθελα να πω ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η προσβασιμότητα θα πρέπει να είναι συνεπής με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ακούσαμε σήμερα για την προσβασιμότητα στο σελίδο δημοσίων φορέων και είναι πολύ σημαντικό να συνδυαστούν οι δύο νομοθετικές πράξεις για να μην δημιουργηθούν ε, προβλήματα. Επίσης, σε σχέση με την οδηγία για τα οπτικαστικά μέσα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η φετινή ε, αναθεώρηση. Αναμένω το έργο που έχουμε μπροστά μας και ελπίζω μέσω των εργασιών και των προσπαθειών που θα καταβάλουμε να καταφέρουμε να κάνουμε τη διαφορά για τους Ευρωπαίους πολίτες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, ε, διεξοδική παρουσίαση του έργου και για την παρουσίαση ε, το συμφωνώ απόλυτα ε, και με αυτό που είπατε για ότι πρόκειται περί πολύ έμπειρου εισηγητή. Συμφωνώ με τα περισσότερα που ανέφερε. Δεν θέλω λοιπόν να επαναλάβω τα ίδια. Να επικεντρωθώ λίγο στις ερωτήσεις μάλλον που μου δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. Ε, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό το νομοθέτημα αυτό που έχουμε μπροστά μας. Ε, και έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε. Αλλά θα πρέπει να αποκόμισουμε και διδάγματα από τις ε, εργασίες σε σχέση με την προσβασιμότητα των ιστοσελίδων. Είναι ένα πολύπλοκο έργο αλλά όχι τόσο πολύπλοκο όσο η προσβασιμότητα στην οποία αναφερόμαστε εδώ. Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη το ότι θα πρέπει να προσεγγίσουμε τις θέσεις Συμβουλίου και Κοινοβουλίου ώστε να βρούμε κοινέ θέσεις ε, και το όλο κείμενο να μην είναι υπερβολικά περίπλοκο γιατί αυτό που αναμένουν από εμάς οι ανάπηροι αλλά όχι μόνο αυτοί, όλοι οι άνθρωποι προς τους οποίους προορίζεται αυτή η νομοθεσία αναμένουν από εμάς ε, το αποτέλεσμα να εμφανιστεί, να είναι ορατό ε, εντό εύλογου χρονικού διαστήματος. Εγώ είμαι λοιπόν υπέρ του να έχει ολοκληρωθεί ε, όλη αυτή η δουλειά σχετικά γρήγορα. Τώρα ερώτηση προς την Κομισιόν. Η Κομισιόν ποια θεωρεί ότι είναι τα σημαντικότερα προβλήματα ε, βάσει των όσων ακούει από το Συμβούλιο τώρα. Και η δεύτερη μου ερώτηση, το άρθρο 12 αναφέρεται στο ανέπαρκες άχθος. Ε, πώς θα το διευκρινίσουμε αυτή την διάταξη ώστε να μην είναι δυνατό, δυνατή η παράκαμψη των κανόνων που έχουν οριστεί. Ε, ο ίδιος φόβος ε, εμφανίζεται όταν μιλάμε για τη λειτουργικό ορισμό της προσβασιμότητας διότι εκεί τα αποτελέσματα δεν αποκλείται να είναι αρκετά σαφή ένας ορισμός ε, που δεν είναι αρκετά περιοριστικός ε, παρέχει ευελιξία σε ο, που μπορεί να συμμορφωθούν με τα κριτήρια αυτά. Αλλά εγώ προβλέπω και επιπλοκές ε, στο έργο αυτό, αλλά όπως είπα από την αρχή, θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντική αυτή η νομοθεσία που όλες μας οι δυνάμεις πρέπει να επικεντρωθούν ε, στους ανθρώπους που θα υποφεληθούν από αυτή την νομοθεσία. Ε, και χαίρομαι ιδιαίτερα για τη συνεργασία μεταξύ μας. Ευχαριστώ. E Ο σκηνόδης των του ECR δεν είναι εδώ. Νταν, έχεις το λόγο. Εκ Ευχαριστώ. Εμείς ε, υποστηρίζουμε το σκοπό της πρότασης, Ωστόσο έχουμε ανησυχίες για το πεδίο εφαρμογή και ιδιαίτερα την μελέτη επιπτώσεων που αιτιολογεί την έκθεση αυτή. Σε σχέση με αυτό που είπε η Κομισιόν ότι συνέταξε με προσοχή τη συγκεκριμένη έκθεση, εγώ πρέπει να διαφωνήσω. Ε, ας είμαστε σαφείς. Πρόκειται για μια μελέτη επιπτώσεων από το 2013 με στοιχεία ακόμη παλαιότερα που μάλιστα απερίφθη από το αρχικό συμβούλιο για την εκπόνησή του και εξετάζει μόνο συγκεκριμένα κράτη-μέλη, ε, μπερδεύει προϊόντα και υπηρεσίες, δεν κατανοεί ακριβώς πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες και δεν καταλαβαίνω ε, για ποιο λόγο θα πρέπει να θεωρηθεί αυτό καλύτερη νομοθεσία, γιατί στην πραγματικότητα ε, πρόκειται για στοιχεία του 2013. Έχουν περάσει ήδη τρία χρόνια στην ψηφιακή εποχή, πρόκειται για μια ολόκληρη γενιά. Ε, νομίζω δηλαδή ότι η Κομισιόν πρέπει ή να επικυροποιήσει τη μελέτη επιπτώσεων ή να εκπονήσει νέα. Και νομίζω ότι η Επιτροπή ΙΜΚΟ θα πρέπει επίσης να ζητήσει και από την υπηρεσία ή PRS του Κοινοβουλίου να εκπονήσει μια τέτοια μελέτη επιπτώσεων. Γιατί πρέπει πραγματικά να ξέρουμε ποιες θα είναι επιπτώσεις. Γιατί διαφορετικά παρά τις θετικές και καλές μας προσθέσεις, προθέσεις θα επιβαρύνουμε τις επιχειρήσεις. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να ε, εξαιρεθούν οι δημόσιες συμβάσεις, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, και νομίζω ότι τα, οι απαιτήσει ε, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν εκείνες που υπάρχουν ήδη στην κλαδική νομοθεσία. Άρα, έχουμε μεγάλο δρόμο μπροστά μας, πρέπει να ξεκινήσουμε από μια νέα μελέτη επιπτώσεων και το λέω αυτό επαναλαμβάνοντας ότι βεβαίως και συμφωνούμε με, ε, τον σκοπό, με τον στόχο αυτής της νομοθεσίας, αλλά έχουμε σοβαρές ε, ανησυχίες και προβληματισμούς σε σχέση με την συγκεκριμένη πρόταση που έχει υποβληθεί. Κύριε Σόλτης. Eh, Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την, εκπρόσωπη, την εκπρόσωπο του, της Κομισιόν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν την Κομισιόν για την πρόταση που έχει υποβάλει. Περιμένουμε αυτή την πρόταση εδώ και αρκετό καιρό. Κάποιοι μάλιστα ισχυρίζονται ότι η πρόταση αυτή δεν είναι αρκετά φιλόδοξη, ότι δεν επιλύει το ζήτημα της ε, προσβασιμότητας στο σύνολό του. Παρόλα αυτά είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την αντιμετώπιση των ε, θεμάτων αυτών. Επίσης Υπάρχουν και διάφορες ε, νομικές ε, πράξεις που ισχύουν σε όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει εμείς να εξασφαλίσουμε την προσβασιμότητα σε προϊόντα και υπηρεσίες για όλους. Και αυτός είναι και ο βασικός στόχος της συγκεκριμένης οδηγίας. Συμφωνώ και με τον ε, συνάδελφο που μίλησε πριν από μένα. Η μελέτη επιπτώσεων θα πρέπει να είναι η βάση για τα πάντα γιατί έτσι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε βιώσιμες λύσεις οι οποίες θα μπορούν και να εφαρμοστούν στο μέλλον. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις που θα επιφέρει συγκεκριμένη πρόταση. Η προσωπική μου γνώμη είναι λοιπόν ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξασφαλίσει ότι δεν θα, δεν θα επιβαρυνθούν υπερβολικά Ιδίω οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να προλάβουμε διάφορα τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να ανακύψουν και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι η Κομισιόν θα πρέπει να προετοιμάσει πρακτικές λύσεις, πρακτικούς μηχανισμούς τους οποίους και θα μπορέσουμε να συζητήσουμε. Και στη βάση αυτών των λύσεων θα μπορέσουμε να ε, επεξεργαστούμε το από εδώ και στο εξή έργο μας. Θα ήθελε κανείς άλλο το λόγο, ρωτάει η Πρόεδρος. Ωραία. Θα ήθελα εγώ να κάνω κάποια σχόλια, αν μου επιτρέπετε. Προσβασιμότητα σε ψηφιακό περιβάλλον είναι απόλυτα σημαντικό θέμα για να ε, ε, δημιουργήσουμε προσβασιμότητα και στον ε, φυσικό κόσμο. Πρέπει να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα λοιπόν και στον εικονικό και στον φυσικό κόσμο. Παρόλα αυτά, όσο περισσότερο διαβάζω αυτήν την πρόταση και όσο περισσότερο τη συζητώ, ανησυχώ όλο και περισσότερο για το ότι αυτή η πρόταση ενδεχομένως να μην είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Αν εξετάσουμε την ομοθεσία για το ψηφιακό περιβάλλον, μιλούμε ε, συνεχώς ότι ε, η καινοτομία ε, κινείται πολύ γρήγορα και θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι οι κανόνες που θεσπίζουμε σήμερα θα μπορούν να εφαρμοστούν και στο μέλλον. Τι συζητούμε εδώ λοιπόν, μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων. Ναι, πριν από κάποια χρόνια μπορεί και να γινόταν αυτό, να πήγαινε σε μηχανήματα έκδοση εισιτηρίων, αλλά τώρα πλέον ε, πα στην εφαρμογή στο κινητό σου, το κατεβάζει το εισιτήριο και δεν χρειάζεσαι καν ε, μηχάνημα έκδοση εισιτηρίων. Για ποιο λόγο εμεί λοιπόν να θεσπίσουμε νομοθεσία η οποία θα ισχύσει και μετά από έξι χρόνια για πράγματα τα οποία δεν θα υπάρχουν κατά πάσα πιθανότητα πια. Ξέρω ότι η Κομισιόν προσπάθησε να είναι πολύ στοχευμένη στις πράξεις της και στις προτάσεις της, αλλά εγώ δεν καταφέρα να καταλάβω πώς ακριβώς χειρίζεστε τους διάφορους κλάδους. Είναι τόσο πολλοί οι κλάδοι που τελικά δεν μου δίνεται η αίσθηση ότι η πρότασή σας είναι σαφής για το τι πρέπει να γίνει. Πράγματι, η μελέτη επιπτώσεών σας βασίζεται σε πολύ παλιά στοιχεία, γιατί, για παράδειγμα, ε, ε, προκύπτει και από διάφορα στοιχεία της ίδιας της, της έκθεσης που έχετε υποβάλει. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για το ποιο θα είναι το κόστος της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων. Ξέρουμε όμως ότι θα υπάρξει κόστος. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Θέλουμε λοιπόν Άνα προϊόν και άνα κλάδο να ξέρουμε τι ακριβώς έχετε ε, χρησιμοποιήσει και συνυπολογίσει ως βάση για να ξέρουμε και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις. Η άλλη ανησυχία που έχω είναι το εξής. Χρησιμοποιούμε πράγματι τα κατάλληλα νομοθετικά εργαλεία Το νέο νομοθετικό ε, πλαίσιο, στο οποίο εγώ έχω εργαστεί ήδη σε, ένα θέμα που αματέθηκε και άλλοι συνάδελφοι, ε, λειτουργεί πολύ καλά για τα αγαθά. Αλλά αυτό δεν δεν σημαίνει ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις την επισήμανση ή την παρακολούθηση της αγοράς για ιστοσελίδες. Δεν τα έχουμε χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαλεία ποτέ. Και φοβάμαι ότι η προσέγγιση ε, όπως, αυτή που είχαμε στην επισήμανση CE δεν είναι πολύ ε, μακρόπνοη. Δεν την έχουμε δοκιμάσει ποτέ στον ψηφιακό κόσμο. Είναι λοιπόν η σωστή βάση. Να πούμε ότι θέλουμε να μεταφέρουμε την επισήμανση CE που αφορά την ασφάλεια των προϊόντων καταναλωτικών αγαθών και να πούμε ότι θέλουμε αυτό το σήμα CE να το βάζουμε και σε ψηφιακές υπηρεσίες. Εγώ ξέρω ότι αυτό το σήμα CE δεν εξελίσσεται και πολύ γρήγορα. Και αυτό είναι καλό γιατί στον τομέα στον οποίο έχει χρησιμοποιηθεί δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη. Εν πάση περιπτώσει, εγώ υποστηρίζω ότι είναι απόλυτη ανάγκη να υπάρχει προσβασιμότητα στον ψηφιακό κόσμο, αλλά δεν έχω πιστεί καθόλου ε, από την μελέτη επιπτώσεων ότι η πρόταση απευθύνεται με το σωστό τρόπο στους κλάδους και στα προϊόντα. Θα ήθελα δηλαδή να σας καλέσω να κάνετε περισσότερες προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα. Ρόμπερτ, ε, θέλεις να απαντήσεις τα όσα ακούστηκαν ή να δώσω το λόγο στην Κομισιόν. Όχι, ο μακρηγόρησα ήδη πολύ, αλλά θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που ήδη βούτυξαν σε αυτό το έγγραφο, πράγμα που αποδεικνύει ότι είναι πολύ σημαντικό για μας. Ε, Έχουμε θέσεις που δεν είναι και τόσο μακριά η μία από Ε, θα δουλέψουμε λοιπόν, θα συνεργαστούμε. Δεν ξέρω αν η Κομισιόν όμως έχει κάποιες απαντήσεις για αυτά τα ερωτήματα που ήδη θέσαμε. <laughs> Come back in, Commission. Thank you. I will μπορείτε να πάρετε το λόγο. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να απαντήσω όσο γίνεται σε περισσότερες από τις ερωτήσεις. Βεβαίω, είναι μια πρόταση που χρειάζεται περισσότερη συζήτηση, όχι μόνο αυτή τη σημερινή και σίγουρα θα πρέπει να επανέλθουμε σε κάποια από τα ε, θέματα που αναφέρατε. Πάντως, ε, κατά τη γνώμη μου, καλύτερη ερώτηση πώς επελέγησαν οι τομείς. Αυτό έγινε με βάση της αξιολογηση αντικτυπου αντικτύπου. Δηλαδή ήταν ε, αρκετά περίπλοκη δουλειά, ε, βήμα-βήμα. Είναι στη σελίδα 15. Ξεκίνησε με τον εντοπισμό πιθανών τομέων που καλύπτονται από τη σύμβαση του ΟΗΕ και ήρθαμε, ε, καταλήξαμε σε ένα κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών που θα μπορούσαν να ε, εμπίπτουν σε αυτή την να καλύπτονται από αυτή την οδηγία. Μετά Είδαμε τις, ε, τη δημόσια διαβούλευση για το ποια προϊόντα θεωρούνται πιο σημαντικά. Επόμενο βήμα ήταν η ιεράρχηση και επιλογή αγαθών και υπηρεσιών που σημαίνει ποιοτική και, και ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο με βάση της, ε, τη δημόσια διαβούλευση για να δούμε πού υπήρχαν αποκλίνουσες απαιτήσει. Αυτή ήταν λοιπόν όπως σας είπα πρώτα η ιεράρχηση αυτή τελειοποιήθηκε με μια κατάλληλη ανάλυση. Και μετά αυτή η ανάλυση εξέτασε τις διάφορες προσεγγίσεις, τις ε, απαιτήσει προσβασιμότητας και με αυτή την τελευταία εις βάθος ανάλυση καταλήξαμε στον τελικό κατάλογο αγαθών και προϊόντων και υπηρεσιών. Και υπάρχουν διάφορα παρατήματα που εξηγούν ε, αυτή την σταδιακή προσέγγιση ώσπου να καταλήξουμε στον τελικό κατάλογο αγαθών και υπηρεσιών. Υπήρχε έπειτα μια ερώτηση για το ρόλο των ε, αρχών εποπτείας της αγοράς που πρέπει να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση ε, των ελέγχων. Ε, θεωρούμε ότι είμαστε σε μια καλή κατάσταση για να το κάνουμε αυτό. Έχουν τις υποδομές και τις μεθόδους και εμείς έχουμε χρησιμοποιήσει ένα νέο νομοθετικό ε, σχέδιο, Βεβαίως αυτό θα απαιτήσει να ε, να τελειοποιήσουμε τις ε, δυνατότητες προσβασιμότητας ε, και εναρμόνισης όταν θα είναι να εγκριθεί αυτή η πρόταση. Έχουμε προβλέψει δύο χρόνια για τη μεταγραφή και τέσσερα χρόνια για την εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής. Θεωρήσαμε ότι ήταν απαραίτητο να έχει χρόνο ο κλάδος αλλά και η ενδιαφερόμενοι να προσαρμοστούν. Ε, λάβαμε υπόψη τα προϊόντα, αλλά και βέβαια όπως είπατε και τους καταναλωτές που θέλουν οπωσδήποτε να ωφεληθούν ή όχι, ή από, αυτές, από αυτό το νομοθέτημα. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι μια ισορροπημένη απόφαση θα ήταν τα έξι χρόνια σύνολο μέχρι ότου εφαρμοστεί η οδηγία και η πρώτη έκθεση να ακολουθήσει ε, μετά από αυτά τα πρώτα έξι χρόνια. Εδώ ε, η επόμενη ερώτηση αφορούσε το περιβάλλον στο οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες. Ε, θεωρήσαμε πως τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποφασίσουν αν και που το, μάλλον κατά πόσο το περιβάλλον όπου δίνονται ή παρέχονται οι υπηρεσίες θα πρέπει επίσης και εκεί να έχουν προσβασιμότητα ή όχι. Η άλλη παρατήρηση ήταν πώς θα εξασφαλίσει η καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην ευθύνη του οικονομικού φορέα και των ε, αγορών, των, μάλλον των αρχών εποπτείας της αγοράς. Αυτό είναι σημαντικό καθώς ε, οι εξελίξεις στον τομέα της πληροφορικής είναι πολύ γρήγορες και θέλουμε να είμαστε σε κάποιο γενικότερο επίπεδο, να μην μπούμε σε ιδιαίτερα με πολλές λεπτομέρειες, ώστε να μην δημιουργήσουμε στενό κορσέ, γιατί οι εξελίξεις είναι πολύ γρήγορες και αν οι λειτουργικές ε, ε, διατάξεις περί προσβασιμότητας μπορεί να περιορίσουν ε, την ανάπτυξη και αυτό δεν το επιθυμούμε. ρωτήσατε ποια είναι η κατάσταση στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο άρχισε να συζητάει αυτήν την πρόταση στα τέλη του Ιανουαρίου. Είχαμε διάφορες συζητήσεις έκτοτε. Οικονομικός αντίκτυπος για την βιομηχανία κυρίως για τις μικρομεσαίες, αλλά υπάρχουν σε αυτό το στάδιο και πολλά πρακτικά ερωτήματα, πρακτικά παραδείγματα. Αν μπείτε στις λεπτομέρειες ε, στα άρθρα θα δείτε ότι χρειάζεται να συζητηθούν ε, διάφορα άρθρα σε λεπτομέρειες και επίσης στα κράτη-μέρη ε, το συζητούν με τους διοικητικούς τους μηχανισμούς, διότι χρειάζεται συζήτηση ανάμεσα σε διαφορετικά υπουργεία σε κάθε χώρα. Υπήρξε και μια ερώτηση για το, την αξιολόγηση αντικτύπου. Εγώ θα παραμείνω στα όσα είπα ότι έχει συνταχθεί πολύ προσεκτικά, ότι ήταν μια πολύ σοβαρή δουλειά που έγινε ε, Και το πιο σημαντικό στοιχείο που προκύπτει είναι ότι μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερος κατακαιρματισμός που σημαίνει περισσότερο κόστος ενώ εμείς θέλουμε να επιτύχουμε καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς καλύτερες ευκαιρίες των βιομηχανιών να ανταγωνιστούν σε ολόκληρη την Ένωση και επίσης ε, έτσι ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να ωφεληθεί από μια ορθώς λειτουργούσα εσωτερική αγορά. Είχαμε κάποια λίγα σχόλια και έπρεπε να το υποβάλουμε δεύτερη φορά. Είναι τώρα όμως ολοκληρωμένη η εξολόγηση αντικτύπου, την έχουμε εγκρίνει και γι' αυτό και θεωρούμε ότι θα έχουμε ξεκινήσει όπως προβλέπετε ε, την ε, σωστή διαβούλευση, όπως προβλέπετε λοιπόν και από τους ε, κανόνες για την καλύτερη νομοθεσία. Περιγράφουμε και με κάθε λεπτομέρεια τα σχόλια που λάβαμε. μετά από την έγκριση του πρότασης ε, οδηγίας. Τέλος, το η σήμανση CE της ε, Ένωσης δηλαδή. Εδώ έχουμε μία πρόταση για ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να έχουμε συνεπή και ε, ταυτόχρονη προσέγγιση σε όλη την πρόταση. Απλά κοιτάω τώρα να δω πώς κάτι ξέχασα. Όχι, εντάξει. Ευχαριστώ. Okay. Thank you very much. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Θα σταματήσουμε για σήμερα και θα συνεχίσουμε αύριο το πρωί στις 9. Να σας προειδοποιήσω και να υπενθυμίσω ότι οι ψηφοφορίες αύριο θα είναι περίπλοκες. Θα υπάρχουν πολλές, γι' αυτό παρακαλώ να είστε όλοι εδώ και να είστε υπομονητικοί. Θα είναι πολύ περίπλοκο το έργο μας αύριο.